So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde dann gerne... Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να κάνω μερικές ανακοινώσεις από τις συνεδρίαση των συντονιστών. Θα μας πάρει λίγη ώρα, οπότε μάλλον θα γεμίσει και η αίθουσα στο μεταξύ. Εχθές αποφασίσαμε τα εξής στις συνεδρίες των συντονιστών. Καταρχάς, η έκθεση του κυρίου Μαστέλα, η κυρία Λίχτεμπεργκερ είναι η συγγητρία. μετά για τη συλλογική διαχείριση. Δεν έχουμε ακόμα να θέσει ε, την έκθεση σε κάποιον εισηγητή. Θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Στι 3 υπάρχει ειδική συνεδρίαση των συντονιστών. Ελπίζω να μην ε, καθυστερήσει πολύ. πέντε λεπτάκια. Στη συνέχεια, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, γνωμοδότηση, την οποία θα συντάξει η κυρία Κάστεξ. τα τα της επίλυσης διαφορών ε, των επενδυτών. Ε, έχουμε αποφασίσει να αναθέσουμε σε εξωτερικό εισηγητή, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Εφαρμογή το οδηγίες ε, για τις υπηρεσίες στα οπτικοακουστικά μέσα. Κάποιο από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, αλλά δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς, θα μάθουμε τον αργότερα, Αναπτυξιακέ πτυχές για τα πνευματικά δικαιώματα, εντάκτη τη νομοδότηση, η κυρία Κάστεξ. Επίσης, συμφωνήθηκε να ετοιμάσουμε και μια γνωμοδότηση για την έκθεση της ΣΥΜΚΟ, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την διακυβέρνηση της αγοράς. Θέλαμε και έγκριση για μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, για τις ε, προσφορές εξαγοράς. Θα είμαι εγώ εισηγητής, αν γίνει αποδεκτή η αίτηση. Κατόπιν έχουμε ένα παρατηρη... Ε, έναν ε, ε, μέλος στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και εγκρίθηκε και μια προφορική ερώτηση για τη σύμβαση της Χάγης για τις απαγωγές παιδιών. Ε, από την κυρία Λίχτεμπεργκερ η προφορική ερώτηση. Είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα γιατί δεν είχε γίνει επίσημη διαβούλευση με τη γραμματεία μας ακόμα. Επίσης θέλουμε να κάνουμε μια συγκριτική ανάλυση για την πρόσβαση σε έγγραφα δικαστηρίου σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια θα αποσταλεί και μια επιστολή προς τον πρόεδρο Σούλτς για τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Παγκόσμιο Φόρουμ ε, Δικαιοσύνης ε, και Ανάπτυξης. Έχουμε επίσης αποφασίσει ότι θα παρουσιαστούν οι απόψεις της ομάδας επικοινωνίας και από με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ε, θα αναθέσουμε μία μελέτη η οποία θα εξετάσει τις περαιτέρω δυνατότητες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επίσης, επιθυμούμε να οργανώσουμε μία ακρόαση που θα αφορά στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού ε, ε, Ιδρύματος. Αυτά έχω να σας πω. Και τώρα, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι συμφωνείτε. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 15. Πρόκειται για το εργαστήριο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων. Ε, γνωρίζετε ότι ε, φέτος υπήρξαν πάρα πολλές ε, ομάδες εργασίας. Αυτή είναι η τελευταία ομάδα εργασίας και θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Βέντα από τη Βιέννη και τον κύριο Βακέα από το Πανεπιστήμιο Λάιντα. Ελπίζω να το πρόφερα σωστά. Σωστά Λάιντα το λέτε. Λάιντα στην Ισπανία. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο και στους δύο εμπειρογνώμονες, να τους δώσω τη δυνατότητα να μιλήσουν ε, και οι δύο συγητέ είναι παρόντες και μετά θα συζητήσουμε και εμείς ε, τις δικές σας τις απόψεις και θα προχωρήσουμε. Νομίζω ε, η κυρία καθηγήτρια μπορεί να ξεκινήσει. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ καταρχάς που μου δίνετε τη δυνατότητα να επισημάνω κάποια ζητήματα τα οποία ε, είχαμε στο ενημερωτικό έγγραφο για τις επιστροφές για το Ευρωπαϊκό ε, Δίκαιο Πολίσεων. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, θα σταθώ σε μερικά βασικά ζητήματα. Κάποια εξ αυτών είναι, καταρχάς, τι είναι αυτές οι επιστροφές, ποιο είναι το περιεχόμενό τους και υπό ποια μορφή θα γίνουν αυτές οι αποδόσεις. Όταν αναφερόμαστε σε αποδόσεις, αυτό το οποίο μας έρχεται κατά νου είναι το κεφάλαιο 17 το οποίο είναι η τελική απόδοση. Και αυτό δεν αφορά μόνο την αποφυγή ή την τελεσίδικη απόφαση. Αν λάβουμε υπόψη μας βέβαια το κεφάλαιο αυτό θα δούμε ότι δεν είναι το μόνο τμήμα το οποίο από λειτουργικής πλευράς αφορά την απόδοση, αλλά ε, στα άρθρα 44 47 έχουμε απόδοση επειδή ο καταναλωτής ε, ε, αποσύρεται από την περιοχή της ε, στην οποία ε, έχει κάνει την καταγγελία και έχουμε και διάφορες άλλες περιπτώσεις. Το κεφάλαιο 17 για την απόδοση, αν το εξετάσουμε στο πλαίσιο των άλλων άρθρων που έχουμε για την απόδοση, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά στο περιεχόμενο αλλά και στη μορφή. έχουμε την προσέγγιση του κεκτημένου της, ε, στα θέματα της απόσυρσης, ενώ στο κεφάλαιο 17 έχουμε ε, μία προσέγγιση 19, αστικού δικαίου του 19ου αιώνα. Δεν Βέβαια αυτό είναι λογικό γιατί η απόσυρση εξαρτάται από το κεκτημένο, βασίζεται στο κεκτημένο. Το κεφάλαιο λοιπόν για την απόδοση αφορά τον πλειονότητα αυτά των περιπτώσεων που προκύπτουν στις ε, ε, συνολικές συναλλαγές. Έχουμε απλούς κανόνες οι οποίοι δεν κατά ανάγκη κομψοί και περιλαμβάνουν και ε, καλά αποτελέσματα τα οποία ως στόχο έχουν να μειώσουν το κόστος των, της επίλυσης διαφορών. Βέβαια μπορεί να μην έχουμε καλή απόφαση σε κάποιες εκ των περιστώσεων αλλά δεν είναι αυτός ο τελικός του στόχος. Αφετέρου, αυτό το οποίο αποκαλώ προσέγγιση αστικού κώδικα 19ου αιώνα είναι θέματα τα οποία αφορούν ε, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ε, διάφορες μορφές δαπανών και δεν αντιμετωπίζουν κάποιες ε, σημαντικές λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα τρόπο με τον οποίο θα γίνει η απόδοση, περιλαμβάνει και λεπτομέρειες όπως ε, σε περίπτωση που ένα αγαθό πρέπει να απεγκατασταθεί από εκεί που το έχουμε εγκαταστήσει. Εδώ γίνεται μια προσέγγιση που δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επίλυσης διαφορών ή άλλο κόστος που μπορεί να προκύψει από αυτή την περίπτωση. Τι πρέπει να γίνει τώρα με τα κεφάλαια αυτά της απόδοσης ε, τι γίνεται τώρα με το ενιαίο κοινοτικό δίκαιο σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει το ενιαίο κοινοτικό δίκαιο να ακολουθεί την ε, ε, προσέγγιση του κεκτημένου ε, και να γραφεί το ενιαίο κοινοτικό δίκαιο προς αυτή την κατεύθυνση σε όλες τις οδηγίες που έχουμε. Καλό θα ήταν όμως να ξαναγράψουμε τουλάχιστον το κεφάλαιο 17 σε σχέση με τα άρθρα 44 έως 47 και το 112 ώστε να θεωρήσουμε ως εφαλτήριο αυτά τα άρθρα και να τα προσαρμόσουμε στο συγκεκριμένο ε, ε, πλαίσιο της ακύρωσης και της καταγγελίας. Και γιατί αυτό, γιατί το κεφάλαιο αυτό στην αρχική του μορφή, αυτό το οποίο σας αποκάλεσα ότι έχει μία προσέγγιση αστικού δικαίου 19ου αιώνα, δεν αντιμετωπίζει κάποια βασικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να αφήσουμε σε κρεμότητα σε ένα νομοθέτημα το οποίο θα εφαρμόζεται σε 27 και άνω ε, διαφορετικές, ε, διαφορετικά νομικά καθεστώτα. Και δεν αντιμετωπίζουμε για παράδειγμα το κατά πόσον ο πολιτής έχει δικαίωμα ή υποχρέωση να δεχτεί τα αγαθά ή αν θα πρέπει να τα ε, παραλάβει ο ίδιος ή αν θα πρέπει ο καταναλωτής να τα αποστείλει, ποιος ε, θα πληρώσει το κόστος της αποστολής, ε, της επιστροφής των αγαθών και επίσης αν χρειαστεί να γίνει η απεγκατάσταση για παράδειγμα έχουμε πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θα ήθελα να σας αναφέρω αυτές τις αποφάσεις αν η υποζημίωση περιλαμβάνει και την παράδοση και σχετικές άλλες δαπάνες και ποιο είναι το εύλογο χρονικό διάστημα για να γίνει ε, η απόδοση. Αυτά όλα ρυθμίζονται στα άρθρα 44-47 και στο 112 και καλό θα ήταν να ε, ρυθμίζονται και στο κεφάλαιο που αφορά στην απόδοση ε, όταν υπάρχει κατά, ακύρωση ή καταγγελία. Αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα και για τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Τώρα, για το ίδιο το κεφάλαιο 17, όπως σας είπα, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, θα πρέπει να περιοριστώ σε τέσσερα βασικά σημεία. Το πρώτο είναι... Η απώλεια η φθορά των αγαθών. Τώρα, ποια είναι η λύση που προκρίνει η πρόταση. Η λύση που προτείνει είναι ο αγοραστής να καταβάλει την νομισματική αξία των αγαθών όταν δεν μπορούν να επιστραφούν καθόλου, αλλά δεν οφείλει καμία πληρωμή σε περίπτωση απλής φθοράς. Τώρα, από συσταλτική άποψη, ε, δεν είναι και πολύ σαφές από το κείμενο της πρότασης, αλλά εγώ τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι ε, κάποια εισαγωγικά κείμενα που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιες δηλώσεις που έκανε και φαντάζομαι ο καθηγητής Στάρτ θα με διορθώσει αν ε, δεν ερμήνευσα σωστά αυτά που διάβασα. Ένας λοιπόν αγοραστής που καλεί την πίστη έλαβε ένα υποκατάστατο ως αντάλλαγμα το, του προϊόντος μπορεί να επιλέξει την επιστροφή, την απόδοση του υποκατάστατου. Αν ε, έχει πωλήσει το αγαθό και έλαβε την τιμή αγοράς ε, πίσω, ο, καλό, ο καλόπιστος αγοραστής μπορεί να επιλέξει να επιστρέψει την ε, τιμή αγοράς που έλαβε από το τρίτο μέρος. Τώρα, για την περίπτωση που ο αγοραστής δεν είναι καλόπιστο, αν δηλαδή ο αγοραστής όφιλε να γνωρίζει τους λόγους ακύρωση ή καταγγελια θα πρέπει, ύστερα από αίτηση του, πολιστή, του πολιτή, να επιστρέψει οποιοδήποτε υποκατάστατο ή την αξία του σε χρήμα. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Καταρχήν, δεν βλέπω την αιτιολόγηση για το ότι, ότι πάντα τον κίνδυνο της απώλειας θα πρέπει να τη φέρει ο αγοραστής και ο πολιτής θα, θα πρέπει πάντα να φέρει τον κίνδυνο της φθοράς. Άσχετα από το ποια ε, ήταν η αιτία της ακύρωσης της καταγγελίας και άσχετα για, το, για ποιο λόγο α, χάθηκαν ή ευθάρισαν τα αγαθά. Επίσης, ε, στην πράξη είναι δύσκολο για ένα δικαστή να τραβήξει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ απώλειας και φθοράς του αγαθού. Για παράδειγμα, ένα καταστραμμένο αυτοκίνητο. Μπορεί κανεί να πει ότι δεν μπορεί να επιστρέψει το αυτοκίνητο γιατί έχει καταστραφεί και ένα καταστραμμένο αυτοκίνητο σαράβαλο δεν είναι πια αυτοκίνητο. Ή μπορεί να το επιστρέψει και να πει ότι έχει φθαρεί. Είναι δύσκολο να γίνει η... να οριστεί διαφορά μεταξύ φθορά και απώλειας. Επίσης, ο, αγορα, ο αγοραστής που έλαβε ως υποκατάστατο 1 ευρώ ε, τη γλιτώνει καταβάλλοντα αυτό το 1 ευρώ. Ενώ ο αγοραστής που δεν έλαβε υποκατάστατο θα πρέπει να καταβάλει την νομισματική του αξία του. Δεν βλέπω τη διαφορά. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η διαφορά, ειδικά όταν πρόκειται για κακόπιστο αγοραστή. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει ο αγοραστής να επιστρέψει το υποκατάστατο αλλά τι γίνεται με την επιστροφή των κερδών, των παράνομων κερδών. Δεν έχουμε όμω επιστροφή παράνομων κερδών σε άλλα σημεία του κοινού δικαίου των ευρωπαϊκών πολίσεων. Τι θα περιμέναμε, για παράδειγμα, στο κεφάλαιο για τι ζημίε ή στο κεφάλαιο για τι επιδόσει. Οπότε το, η επιστροφή των παράνομων κερδών είναι ε, ε, αποδεκτός κανόνας, αλλά στην περίπτωση αυτή είναι ένα ξένο στοιχείο. Ποια θα ήταν η δική μου πρόταση. Η δική μου πρόταση θα ήταν να έχουμε ένα κανόνα που να αναφέρεται στο κεφάλαιο 16 για τις ζημίες, οπότε ο ε, αγοραστής να καταβάλει τις ζημίες αν δεν μπορεί, να επιστρέψει το αγαθό ή αν έχει υποβαθμιστεί το αγαθό. Στο μέτρο όμως που η απαξίωση ξεπερνάει τη φθορά από κανονική, από φυσιολογική χρήση ή δεν υπάρχει σύγκρουση με τους κανόνες ε, της χρήσης. Πάντως γενικός αγοραστής είναι υπεύθυνο, αλλά δεν είναι υπεύθυνο όταν υπάρχει εύλογος λόγος. Επίσης δεν είναι υπεύθυνο το μέτρο που η φθορά ή η απώλεια προκλήθηκαν από τον πολιτή και ιδιαίτερα από το γεγονός ότι τα αγαθά δεν ανταποκρινόταν στο περιεχόμενο της σύμβασης. Είναι επίσης δύσκολη η σχέση μεταξύ των κεφαλαίων των κανόνων της απόδοσης και του κεφαλαίου για τις κανόνες ε, της, ε, των επιδόσεων και της ε, επιστροφής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους καρπούς. Τους καρπούς, τη χρήση και τους τόκους. Φαίνεται ότι ο αγοραστή πρέπει να επιστρέψει οποιουσδήποτε φυσικού ή νομικού καρπούς έχει αποκομίσει, αλλά υπό σαφώ προσδιορισμένε περιπτώσει. Ο πολιτή θα πρέπει να καταβάλει τόκο μόνο όταν ο αγοραστή ε, καταβάλει ένα τίμημα για τη χρήση ή σε περίπτωση απάτη, για παράδειγμα. Και μεταξύ των περιπτώσεων όπου ο αγοραστή πρέπει να πληρώσει για τη χρήση, όπω είναι η περίπτωση που δεδομένη τη φύση του αγαθού, την, ε, τη ζήτηση και τα ένδικα μέσα πέραν της καταγγελίας θα ήταν άδικο να επιτρέψουμε ε, στον αγοραστή την ε, δωρεά χρήση για μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτά προβλέπει ο κανονισμός. Βέβαια, όταν δούμε τις αρχές του ρωμαϊκού δικαίου και θέλουμε να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ των καρπών και της χρήσης, της επικαρπής και τις χρήσεις, ε, εντάξει, αλλά για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ καρπών επικαρπίας και χρήσης. Θα πρέπει να τη χάνουν ίσης μεταχείρισης. Ιδιαίτερα ε, ο κανόνας ότι ο πολιτής θα πρέπει να καταβάλει τόκο μόνο σε σαφώς προσδιορισμένες περιπτώσεις ενώ ο αγοραστής σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιστρέψει τους καρπούς που αποκόπησε, πιστεύω ότι είναι άδικο. Θα πρέπει να τύχουν ίση μεταχείριση και ο πολιτής και ο αγοραστή. Οπότε ο αγοραστή θα πρέπει να επιστρέφει τους καρπούς, επίσης επί στενά προσδιορισμένους όρου που ισχύουν και για τη χρήση και για το στόκους. Ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα είναι ότι ε, ο κανόνας για την περίπτωση, ο κανόνας που θα ήταν άδικο να αφήσουμε στον αγοραστή δωρεάν χρήση. Αυτός ο κανόνας είναι πολύ επικίνδυνος γιατί δημιουργεί ασάφεια και αβεβαιότητα για τα συμβαλόμενα μέρη. Δεν ξέρουν αν ο αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει για τη χρήση μετά την καταγγελία και αυτό κάνει ακριβώς το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων ε, ε, λίγο ελκυστικό και αποτρέπει τους καταναλωτές να ασκήσουν το δικαίωμα της καταγγελίας τους γιατί δεν ξέρουν αν θα πρέπει να καταβάλουν ένα αποτρεπτικό ποσό αποζημίωση και αυτό το γεγονός του αποτρέψει από το να ασκήσουν το δικαίωμα καταγγελία. Εγώ θα προτιμούσα ένα σαφή και πιο ταχύ κανόνα με βάση τον οποίο ο αγοραστή που συνήθω δεν υποχρεώνεται να πληρώσει για την χρήση εκτό και αν ήταν κακόπιστο. και φυσικά αυτό ήταν ένα πολύ φιλικό προ τον αγοραστή κανόνα, που ίσω όμω δημιουργήσει κάποια προβλήματα ε, στου καταναλωτέ αλλά εγώ θα προτιμούσα μία μικρή, ε, ένα μικρό περιορισμό των δικαιωμάτων καταναλωτών στη φάση των ενδίκων μέσων, για παράδειγμα για τα καταναλωτικά ε, ε, συμβόλαια να υπάρχει το δικαίωμα του πολιτή για επιστροφή σε περίπτωση, να μην δεχτεί την επιστροφή σε περίπτωση εξατομικευμένων προϊόντων και επίσης για το εξάμεινο να μην υπάρχει το δικαίωμα αυτό για τον πολιτή, να μην δεχτεί την επιστροφή και μετά ε, να μην υπάρχει ε, δυνατότητα για τον αγοραστή, ε, να μην υπάρχει υποχρέωση του αγοραστή να καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση χρήση. Νομίζω ότι έτσι αυξάνεται το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Επίσης, ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο. Ο κανόνα που ισχύει τώρα είναι ότι ο πελάτη που έλαβε ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να καταβάλει σε κάθε περίπτωση την νομισματική του αξία, άσχετα αν έχει καταβληθεί αυτό το ψηφιακό περιεχόμενο σε υλικό μέσο ή άσχετα με τους λόγους ακύρωση καταγγελίας. Επίσης υπάρχει ο κανόνας που λέει ότι η νομισματική αξία είναι το ποσό που ο καταναλωτής, ίσως θα πρέπει να λέμε ο πελάτης, ε, εξοικονόμησε κάνοντας χρήση του ψηφιακού περιεχομένου. Κατά τη γνώμη μου, η εφαρμογή αυτού του κανόνα είναι πολύ δύσκολη στην πράξη. Επίσης, το υλικό μέσο θα πρέπει να το κρατήσει ο αγοραστής ή θα πρέπει να το αποδώσει, να το επιστρέψει ή ο πελάτης θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το ψηφιακό περιεχόμενο και να ε, πληρώνει ή μπορεί να απόσχει από οποιαδήποτε χρήση του ψηφιακού περιεχομένου στο μέλλον. Και αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να πούμε τι εξοικονόμησε ο πελάτης όταν φορτώνει ένα παιχνίδι, ένα μουσικό κομμάτι, μια ταινία. Είναι δύσκολο να αποτιμήσουμε το τι εξοικονομεί σε τέτοια περίπτωση δεν νομίζω ότι είναι καλός κανόνας να λέμε ότι θα πρέπει ο πελάτης να, καταλά... να καταβάλει την νομισματική αξία ακόμη και αν μπορεί να αποδώσει ένα υλικό μέσο που είναι σφραγισμένο. Δεν θα πρέπει να ισχύει αυτός ο κανόνας για το ψηφιακό περιεχόμενο. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ο πολιτής ψηφιακού περιεχομένου υπόκειται στα διαχειριστικά πλαίσια του ψηφιακού περιεχομένου. Η ακολούθητη λύση φυσικά εξαρτάται από μία απόφαση πολιτικής. Πάντως θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα στις διάφορες περιπτώσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο πελάτης δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει στο μέλλον καθόλου το ψηφιακό περιεχόμενο το θέμα του υλικού μέσου, του υλικού υποθέματο, θα πρέπει να το εξετάσουμε σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό περιεχομένο, αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Θα πρέπει να υιοθετηθεί διαφορετική λύση. Σε ορισμένε περιπτώσει δεν μπορούμε καν να εξακριβώσουμε αν ο πελάτη θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί όχι το ψηφιακό περιεχόμενο. Και έχουμε και την τελευταία περίπτωση που ιδιαίτερα είναι πολύ δύσκολη να ε, λυθεί και θα πρέπει εκεί να ληφθεί μια απόφαση επιπολιτική. Και το τελευταίο θέμα, η ρήτρα ελαστικότητας. Είναι κάτι που επικρίθηκε δρυμαίως. Αναφέρομαι στο άρθρο 176 της πρότασης που προβλέπει ότι οποιαδήποτε υποχρέωση επιστροφής ή πληρωμής σε δυνάμει του κεφαλαίου μπορεί να τροποποιηθεί στο μέτρο που η επίδοση η επίδοση του θα ήταν άδικη, λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι το συμβαλόμενο μέρο δεν προκάλεσε ή δεν αναγνώρισε το λόγο ακύρωση ή καταγγελία ασκήθηκαν δερμήτα τις επικρίσεις για το κανόνα αυτό. Τις αντιλαμβάνομαι αυτές τις κριτικές, γιατί όντως είναι κάπως ασαφής αυτός ο κανόνας για τα συμβαλόμενα μέρη, αλλά σε τελική ανάλυση πιστεύω ότι αυτό είναι το τίμημα που καταβάλει κάποιος όταν υιοθετεί σύντομους και σαφείς κανόνες. Είναι δύσκολο να έχουμε ένα νόμο για τις αποδόσεις, για τις επιστροφές που δεν θα είναι ελαστικός θα πρέπει να τον κρατήσουμε, αλλά η εφαρμογή του να, να ισχύει σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε <clears throat> πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, παρακαλώ, ε, έχετε το λόγο. Good morning. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι αγαπητοί Ευρωβουλευτέ. Εγώ θα περιοριστώ στα πιο ουσιώδη ζητήματα της παραγραφής, κεφάλαιο 18 δηλαδή του κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου Πολίσεων. Σας έχω υποβάλει και εκτενές έγγραφο. Το πρώτο θέμα είναι το πεδίο εφαρμογής του κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου των Πολίσεων, του ΣΕΣΛ. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως δείχνει και ο τίτλος του, αφορά μόνο τις πωλήσει, γιατί πρόκειται για κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πωλήσεων. Υπάρχουν όμως α, ε, ε, κεφάλαια που μιλάνε για τις ε, άδικες, άδικους όρους, για τις διάφορους όρους του συμβάσεων, που εμπίπτουν στις γενικές κανόνες, οποιοδήποτε, στις γενικές διατάξεις οποιοδήποτε αστικού δικαίου. Το θέμα της παραγραφής διαθετείται στο τελευταίο κεφάλαιο του ΣΕΖΛ, στο κεφάλαιο 18, και δεν αναφέρεται πουθενά η διάκριση μεταξύ αγοραστή και πολιτή. Αναφέρονται συμβαλόμενα μέρη, αναφέρονται ε, πρόσωπα, αναφέρεται ο φιλέτης και επιστοτής ή δανειστής, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται πολιτής και αγοραστής στο κεφάλαιο της παραγραφής, στο κεφάλαιο 18. Επίσης, έχουμε μια διάταξη που μιλάει για την παραγραφή σε περίπτωση προσωπικών βλαβών. Ε, οι προσωπικές βλάβες μπορεί να μην σχετίζονται κατά ανάγκη με τις πωλήσει. Τι γίνεται όμως αν οι κανόνες αυτοί εφαρμοστούν σε όλες τις υποχρεώσεις που είτε απορρέουν είτε όχι από ένα πολιτήριο συμβόλαιο. Ή μήπω αυτές θα πρέπει να περιορίζονται ακριβώς στις συγκεκριμένες πωλήσει. Γιατί η παρούσα διάταξη όπως έχει διατυπωθεί δεν δίνει σαφή απάντηση για το ποια λύση προκρίνεται στην περίπτωση αυτή. Ένα άλλο θέμα αφορά το γεγονός ότι αυτό το ΣΕΣΕΛ, το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων, καλύπτει το ΠΕΚΛ ουσιαστικά και το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς, DCRF. Ορισμένες όμως διατάξεις είτε παραλήφθηκαν είτε τροποποιήθηκαν. Και αυτή η τροποποίηση των δικονομικών κανόνων στο σχέδιο του κοινού πλαισίου αναφορά στο DCRF, δεν ήταν πάντα επιτυχής. Γιατί διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στον κανονισμό για το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων. Τώρα η τελευταία γενική ερώτηση αφορά τα προβλήματα με τους ορισμούς. Για παράδειγμα, αναφέρεται κάπου η διαμεσολάβηση. Ουσιαστικά γίνεται μια αντιγραφή της αντίστοιχης οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τη διατησία. Αλλά το θέμα της έναρξης ε, των δικαστικών ε, διαδικασιών, η αναγνώριση, σημαντικές έννοιες ε, όπως η διαπραγμάτευση, το συμπληρωματικό δικαίωμα, ancillary right, δεν προσδιορίζονται σαφώς, κάτι που δημιουργεί ασάφεια και προβλήματα στον ορισμό. Στο ΠΕΚΛ, το αντικείμενο της παραγραφής είναι η αξίωση, η απέτηση. Άσπρουχ, όπως λέμε στα γερμανικά. Είναι η μετάφραση του άσπρουχ, η απέτηση, που είναι το δικαίωμα ουσιαστικά τέλεσης μιας υποχρέωσης. Αυτό λέει και το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων. Απλώς προσθέτει το δικαίωμα επιβολής μιας υποχρέωσης. Της εκτέλεσης δηλαδή μιας υποχρέωσης. Το δικαίωμα να εξαναγκαστεί κάποιος σε εκτέλεση μιας υποχρέωσης. Το άρθρο 184 ή συγγνώμη, το άρθρο 178 δεν αναφέρεται μόνο στο δικαίωμα να ε, ξαναγκαστεί κάποιο εκτέλεση υποχρέωση, αλλά αναφέρεται σε οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαίωμα. Τι θα πει όμω συμπληρωματικό δικαίωμα, ancillary right, μια και δεν προσδιορίζεται αυτό το συναφέ ή επικουρικό ή συμπληρωματικό δικαίωμα. Μία απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι και το συμπληρωματικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα εξαναγκασμού σε εκτέλεση μια υποχρέωση, τη υποχρέωση καταβολή στόχου για παράδειγμα. Αλλά τότε δεν έχει νόημα να πούμε το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση ή οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαίωμα, μια και το συμπληρωματικό δικαίωμα θα είναι το ίδιο. Μια άλλη πιθανότητα είναι το ancillary right, το συμπληρωματικό δικαίωμα, να είναι οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διαφορετικό από αυτό της, το εξαναγκασμού σε εκτέλεση της υποχρέωσης. Οπότε θα καλύπτει ένδικα μέσα όπω η παρακράτηση τη επίδοση, η μείωση τη τιμή ή η καταγγελία τη σύμβαση. Σε ό,τι αφορά την μη ε, εκτέλεση διαβάσουμε το άρθρο 185 παράγραφος 1 βλέπουμε ότι δεν υπόκειται σε καμία παραγραφή. Και αν δούμε το θέμα της μείωσης του τιμήματος, θα μπορούσαμε και αυτό να το εκλάβουμε ως ε, δικαίωμα επιβολής ε, της υποχρέωσης, ε, μια και το δικαίωμα είναι το δικαίωμα να το επιστραφεί ή το υπερβάλλον της τιμής. Οπότε μας μένει μόνο η καταγγελία. Η καταγγελία όμως μερικές φορές εξαρτάται από την έγκαιρη προειδοποίηση. Για παράδειγμα 190-139. 119 συγγνώμη, και 139. Το θέμα είναι αυτός ο έθετος χρόνος, αυτή η έγκαιρη προειδοποίηση. Είναι και ο χρόνος της παραγραφής. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις δεν απαιτείται η ενημέρωση η κοινοποίηση. Για παράδειγμα, στο άρθρο 119.2β και το 139.3 δεν προβλέπεται τέτοιο, τέτοια υποχρέωση ε, κοινοποίηση. Τι γίνεται, η καταγγελία υπόκειται σε παραγραφή, όχι. Οπότε αυτό, αυτή η έννοια του συμπληρωματικού δικαιώματος ή του, παρε, του παρεπόμενου δικαιώματος δεν είναι σίγουρο. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν με τον ορισμό του ancillary right του παρεπόμενου δικαιώματο. Επίση, το θέμα τη περίοδου παραγραφής. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν δύο περίοδοι παραγραφή, Μία σύντομη περίοδο, που είναι διετή και μία πιο μακρά περίοδο, που είναι 10 χρόνια συν 30 χρόνια περίοδο για την περίπτωση προσωπικών βλαβών. Δεν ξέρουμε όμω σε τι αξιώσει, τι απαιτήσει ή τι δικαιώματα εφαρμόζονται αυτέ οι διαφορετικέ περίοδοι παραγραφή γιατί δεν αναφέρεται τίποτα στη διάταξη. Δεν έχει νόημα να έχουμε μια γενική περίοδο παραγραφής. δεν έχει νόημα να έχουμε δύο γενικές περίοδους παραγραφής. Εκτός αν έχουμε μια γενική περίοδο παραγραφής και μια ειδική περίοδο παραγραφής. Αλλά δύο γενικές περίοδοι παραγραφής είναι λίγο παράλογο. Στο DCRF έχουμε μία γενική περίοδο τριετή. Οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η σύντομη περίοδος, η διετής, είναι η γενική. Αλλά σε τι απαιτήσει εφαρμόζεται, σε τι δικαιώματα, ε, για τι δικαιώματα ισχύει η δεκαετής, η πιο μακρόχρονη περίοδος παραγραφής. Μία άλλη πιθανότητα, η εναλλακτική λύση, θα ήταν η δεκαετής περίοδος, να μην είναι περίοδος παραγραφής, αλλά μία μακρά διακοπή, long stop αλλά θα σας αποδείξω αργότερα ότι στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο πολίσεων δεν υπάρχει κανόνας long stop. Γιατί η έναρξη της ε, παραγραφής, σε σχέση με τη σύντομη περίοδο παραγραφής, εξαρτάται από τη γνώση. Είναι η υποκειμενικό λοιπόν το θέμα το πότε, θα, ε, πότε έχει γνώση για, να ενεργοποιηθεί η παραγραφή. Επίσης, ε, αναφέρεται ένας λόγος για την αναστολή της σύμβασης και δύο λόγοι για την αναβολή. Σε ό,τι αφορά την ε, αναστολή, τη διακοπή, έχουμε την αρχή της, των δικαστικών διαδικασιών ως λόγο διακοπής, ε, λόγω αναστολής. Αλλά τι θα πει έναρξη δικαστικών διαδικασιών, μια και δεν υπάρχει ορισμός τη της έναρξης των δικαστικών διαδικασιών, των δικαστικών διαδικασιών δεν ξέρουμε πότε αρχίζουν. Στα περισσότερα δικονομικά συστήματα βέβαια, οι δικαστικές διαδικασίες είναι συνήθως λόγος για ανανέωση της παραγραφής ή για διακοπή της παραγραφής. Το κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων ακολουθεί την πιο σύγχρονη γραμμή και θεωρεί ότι δεν είναι λόγος ε, ε, ανανέωσης, αλλά είναι λόγος ε, αναστολής της παραγραφής η έναρξη των δικαστικών διαδικασιών. Κανένα πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι κάθε είδους δικαστική διαδικασία οδηγεί σε αναστολή της παραγραφής. Για παράδειγμα, διαδικασίες εκτέλεσης που προϋποθέτουν εκτελεστήριο τίτλο του πιστωτή. Επίσης ε, διακόπτουν την παραγραφή ή μήπως υπάρχει ανανέωση της παραγραφής. Ένα άλλο επίμαχο ζήτημα για την αναστολή της παραγραφής και τους λόγους αναστολής της παραγραφής βρίσκεται στο άρθρο 186 ή ε, μάλλον 181 διορθώνει ο μιλητή. Εκεί στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι όταν οι διαδικασίες ε, ε, ε, ολοκληρώνονται πριν το εξάμεινο, χωρίς να εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας, η προθεσμία παραγραφής δεν πριν την πάροδο 6 μηνών από το πέρας της διαδικασίας. Αλλά μπορεί να έχουμε εγκατάλειψη της αγωγής ε, του πιστωτή και έτσι να μην εκδοθεί ε, απόφαση επί της ουσίας. Οπότε γιατί να μην ισχύει και σε περίπτωση που υποβάλλεται η αγωγή σε μία αρμόδιο δικαστήριο. Επίσης γιατί να αναφέρεται η εξάμηνη περίοδος. Και επίση ε, υπάρχει αναβολή, δεν υπάρχει αναστολή, γιατί προβλέπεται ένα επιπλέον εξάμεινο παραγραφής εδώ. Κατά τη γνώμη μου, η, το κόλλημα για λόγους που δεν υπόκειται σε έλεγχο είναι επίσης λόγος για αναστολή. Κάτι που δεν αναφέρεται στο κείμενο. Πιστεύω ότι και αυτό το κόλλημα, αν δεν ευθύνεται ο αγοραστής, θα πρέπει να θεωρηθεί ως λόγος αναστολής παραγραφής. Τώρα, λόγοι της αναβολής που αφορούν την ανικανότητα είναι μονομερείς. Γιατί αφορούν μόνο τον οφηλέτη που δεν έχει εκπρόσωπο. Γιατί όμως θα πρέπει να είναι μονομερείς αυτός ο λόγος και να μην ισχύει διμερός, αμφίδρομα. Γιατί να περιορίζεται μόνο δηλαδή στη μία συμβαλόμενη πλευρά, μόνο στον οφειλέτη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μέγιστη περίοδο, το σημείο 26 του Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου Πολίσεων κάνει μια διάκριση μεταξύ της παραγραφής και της άρσης. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια παράταση στους ε, κανόνες. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, διάταξη για την long stop period. Στο 181 αναφέρονται και οι δύο περίοδοι. Στο άρθρο 182 και 183 αναφέρεται μία περίοδος και το 186 μιλάει για ε, συντόμευση ή επιμήκυση και των δύο περίοδων. Η συντόμευση ή επιμήκυση όμως των περίοδων δεν συμβαδίζουν με τον κανόνα long stop. Και ο κανόνας long stop είναι σημαντικός. Γιατί η έναρξη της, της σύντομης παραγραφής εξαρτάται από τη γνώση. Οπότε, όταν ο πιστωτής δεν έχει γνώση, δεν ξεκινά η παραγραφή. Σε ό,τι αφορά την ανανέωση της περίοδου παραγραφής, η καινοτομία μιας νέας σύντομης περίοδου, σε περίπτωση που διακοπεί η παραγραφή δηλαδή, θα πρέπει να αναθεωρηθεί, να επανεξεταστεί. Για παράδειγμα, τι γίνεται με την αξίωση σε περίπτωση προσωπικών βλαβών, που είναι σχεδόν 30 κοντατή παραγραφή με βάση το ΣΕΣΙΛ. Αν μετά από ένα χρόνο ο φιλέτης αναγνωρίσει την ύπαρξη του δικαιώματος, και λάβει χώρα αυτή η ανανέωση της παραγραφής, η παράταση, τότε έχουμε μόνο τη σύντομη περίοδο, τα δύο χρόνια. Οπότε στην πράξη τριακατοετής περίοδος δεν είναι τριακατοετής στο περίπτωση αυτή. For the, um, Και νομίζω ότι αυτό είναι επιπλέον χρόνο για τον οφηλέτη. Υπάρχει τώρα ένα πρόβλημα όταν αναμειγνύονται τα διάφορα αποτελέσματα. Δηλαδή, το ασθενές αποτέλεσμα ο φιλόετης μπορεί να αρνηθεί την, την εκτέλεση και το δεύτερο είναι το μακροπρόθεσμο, το πιο ισχυρό, ότι πλέον ε, έχουν ε, πάψει να υπάρχουν τα γενεσχουργά αίτια και αυτό είναι λίγο περίεργο γιατί εδώ αναμειγνύουμε τα δύο αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα την αυτονομία των μερών, δεν είναι σαφές για ποιο λόγο έχουμε αυτή την ε, αυτονομία των μερών. Διότι το άρθρο λέει πιο συγκεκριμένα και ξέρουμε ότι αυτό το πιο συγκεκριμένα δίνεται για λόγους έμφασης ή για να μας δώσει κάποιο παράδειγμα. Είναι αμφισβητήσιμο λοιπόν το κατά πόσον τα δύο μέρη μπορούν να μετατρέψουν την περίοδο αναβολή σε περίοδο ανανέωσης ή μπορούν να προσθέσουν νέες λόγους για, για αναστολή ή αναβολή και ούτω καθεξής. Και δημιουργείται μια σύγχυση εδώ, διότι υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι σε μια σύμβαση μεταξύ ενός εμπόρου και ενός καταναλωτή μπορεί να μην εφαρμόζεται εις βάρος του καταναλωτή και αμέσως μετά λέει ότι τα δύο μέρη χαίρουν της μέγιστης δυνατής αυτονομίας και μπορούν να εισαγάγουν αλλαγές και λέει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλησης αυτής της διάταξης από τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Σας επεσήμενα λοιπόν τα πιο διαφιλονικούμενα ζητήματα εδώ, τα πιο επίμαχα και κατά την άποψή μου η διατύπωση του Ευρωπαϊκού Κοινού Δικαίου Πολίσεων δεν είναι ικανοποιητική. Μπορούμε να πούμε ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αλλά η DCFR και η PECL προσφέρουν ένα πιο συνεπές σύστημα κανόνων παραγραφής. και ίσως αν εγκρίνουμε τους κανόνες του DCRF ε, στο σύνολό τους και έχουμε κοινώνες, κοινούς κανόνες για την παραγραφή θα ήταν καλύτερη η λύση σε αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Vielen herzlichen Dank, Herr η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, επομένως θα σταθώ στα σημαντικά. Να ξεκινήσω με την τελευταία φράση του καθηγητή Βάκε, ο οποίος πρότεινε οι κανόνες αυτοί να χρησιμοποιηθούν από το DCRF. Ε, ε θα ήθελα να σταθώ στα βασικά σημεία που είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τι βλέπει, είναι και πολιτικό το ζήτημα και πώς το βλέπουμε εμείς αυτό την προθεσμία αναστολής και την προθεσμία ανανέωσης. Θα πρέπει εδώ να σας παραπέμψω στην οδηγία του 8944 για τις αγορές. Η οδηγία αυτή δεν προβλέπει προθεσμίες παραγραφής, αλλά έχει μία προθεσμία δύο ετών εντός της οποίας θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό φυσικά δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν μια προθεσμία παραγραφής η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο χρόνια από την παράδοση του αγαθού και επομένως ε, τότε εκπνέει και η προθεσμία. Η πλειονότητα λοιπόν των κρατών μελέων έχουν λοιπόν τη συγκεκριμένη προθεσμία και κάποια έχουν προθε... περιορίσει αυτή την προθεσμία. Τι κάναμε λοιπόν εμείς στο δίκαιο πολίσεων, εμείς έχουμε μόνο μία προθεσμία, δηλαδή έναν κανονισμό που ε, συνεπάγεται λιγότερες δαπάνες ε, από τους περισσότερους εθνικούς κανονισμούς. Ε, γιατί εμείς προβλέπουμε μόνο την προθεσμία απόσβευσης και παρετούμεθα από την προθεσμία που έχει σχέση με την, το αντικείμενο της παραγραφής περισσότερο. Η απάντηση είναι απόλυτα σαφής. Στην πρακτική τα δικά μας τα συστήματα έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα από DSFA και PECL ε, που έχουν ε, ένα αντικειμενικό σημείο κίνησης και μετά προσθέτουν μία τριετή χρονική περίοδο. Αυτή η προθεσμία όμως μπορεί να ανασταλεί στην περίπτωση όπου υποθέτει ο ε, αγοραστής ότι υπάρχει κάποιο έλλειμμα. Εδώ η χρονική περίοδος ανέρχεται σε 10 έτη. Άρα δηλαδή καταλήγουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί αν πει κανεί ότι ξεκινάει η προθεσμία από την ε, ημερομηνία παράδοσης και μετά ε, προβλέπεται μίνιμουμ τριετής περίοδο και κατά το μέγιστο δεκαετής, καταλήγουμε στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Δηλαδή έχουμε ένα σύντομο χρονικό διάστημα που ξεκινάει από την υποκειμενική άποψη της ε, υποτιθέμενης γνώσης, αλλά η μέγιστη χρονική περίοδος είναι 10 χρόνια. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι προκύπτουν 2 ε, χρόνια στο σύντομο χρονικό διάστημα, αντί για 3 χρόνια από το DSF. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί επιλέξαμε την υποκειμενική ημερομηνία έναρξης, διότι... Ε, αυτό που υποπτεύεται ως έλλειμμα ο αγοραστής, γι' αυτό υπάρχουν τρία σημαντικά στοιχεία. Ε, το πιο σύγχρονο, η πιο σύγχρονη νομολογία είναι η γαλλική του 2008 και ξεκινάει με ένα υποκειμενικό σημείο κίνησης. Δεύτερον, υπάρχει μια διεθνή στάση και τρίτον, η, ε, το μόνο προηγούμενο που υπάρχει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την παραγραφή και εκεί προβλέπεται μια υποκειμενική ε, προθεσμία αλλά κυρίως η ηλική αν θέλετε εισαγωγικά αιτιολογία είναι ότι επιτρέπεται ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν τα τρία χρόνια που πρότεινε η ομάδα εμπειρογνωμόνων και που ε, συμπεριλαμβάνει και η DSF και PECL. Τα δύο αυτά έτη στις κανονικές συναλλαγές ε, έχουν πλέον συμπεριληφθεί. Δηλαδή όλοι το ξέρουν αυτό τα δύο χρόνια. Και γι' αυτό πλέον και εμείς επιλέξαμε αυτά τα δύο χρόνια όμως ε, από τη στιγμή απόκτησης της γνώσης ή από τη στιγμή που υποπτεύεται ο αγοραστής ότι γνωρίζει. Η DSRF ε, και ΠΕΚΛ ε, επέλεξαν υποκειμενικά μία μακρά περίοδο. Γιατί τι λένε, ότι μπορεί ο αγοραστής να μην μάθει ποτέ ή να μην υποπτευτεί ποτέ. Σπάνιο, αλλά υπάρχει. Και χρειάζεται, εν να υπάρχει μια καταληκτική περίοδος. Αυτά τα δέκα έτη πράγματι συνεπάγονται νομική ασφάλεια. Τώρα, όσον αφορά τα δέκα χρόνια. Τα δέκα χρόνια ε, υπερτιμούνται στη συζήτηση. Γιατί διότι πολύ συχνά αναφέρεται ότι μα ο αγοραστής είχε 10 ολόκληρα χρόνια για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Στην πράξη όμως αυτό δεν ισχύει και θα σας πω γιατί. Πρώτον, διότι η υποκειμενική προθεσμία όσο τρέχει αυτή δεν τρέχουν παράλληλα τα 10 έτη και αυτό αναφέρεται στο άρθρο 185 που αναφέρει ότι όταν ε, καταπίπτει μία ημερομηνία καταπίπτουν όλες οι άλλες, δηλαδή προκύπτει παραγραφή. Άρθρο 185, άρθρο 1, εκεί αναφέρεται ότι δεν ισχύει πλέον η μακρά περίοδος, άρα ισχύουν τα δύο χρόνια. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οι έναρξη των δύο ετών δεν ξεκινάνε από την απόκτηση της γνώσης, αλλά και καθαρά από την υποψία όπου ο αγοραστής ε, θα έπρεπε να υποπτεύεται ή να γνωρίζει. Στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι τέτοιο συμβαίνει πολύ νωρίτερα, δηλαδή ε, αν θέλετε έξι εβδομάδες μετά την παράδοση όταν χρησιμοποιεί κανείς το αντικείμενο. Ε, πολύ σπάνια, σε πραγματικά εξαιρετικές περιπτώσεις εμφανίζεται αυτό το θέμα αργότερα. Άρα δηλαδή στην πράξη μιλάμε για δύο χρόνια από την ε, ύπαρξη υποψίας και τα δύο χρόνια δεν έχουν καμία σχέση με τα δέκα. Το δεύτερο που θέλω να πω και είναι εξίσου σημαντικό είναι το εξής. Ας υποθέσουμε χάρη της επιχειρηματολογίας το λέω αυτό. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο αγοραστής ε, γνωρίζει την, ε, το πρόβλημα, την έλλειψη μετά από 10 χρόνια. Σπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει χάρη του επιχειρήματος ας το πούμε ότι υπάρχει αυτή η υποψία ελαττώματος και έτσι λοιπόν ας υποθέσουμε πράγματι ότι το ελάττωμα υπήρχε πράγματι πριν από 8 ολόκληρα χρόνια. Δεν συμβαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα δηλαδή τα 10 χρόνια έχουν πολύ μικρότερη σημασία από ότι στην πολιτική συζήτηση. Αυτά τα 10 χρόνια ε, χρησιμοποιούνται μόνο και μόνο για να υπάρξει νομική ασφάλεια. Έχει περάσει πάρα πολύ ώρα, αλλά παρόλα αυτά θα κάνω δύο παρατηρήσεις ε, σχετικά με την ε, ομιλία της κυρίας Βέντεχόρστ. Η κυρία Βέντεχόρστ ε, επέκρινε ορισμένα σημαντικά θέματα και επέκρινε το τι υπάρχει στο άρθρο, συγγνώμη, μιλητής, διορθώνω, στο κεφάλαιο 17, στο μοντέλο της απόδοσης. Εδώ ε, υπάρχουν μόνο δύο θέματα και θέλω να σας εξηγήσω γιατί ε, επιλέξαμε αυτή τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Δικαίου Πώλησης ε, παρότι βέβαια κανείς δεν αμφισβητεί την ουσία. Εν περιπτώσει, σε επίπεδο αρχής έχουμε δύο διαφορετικά μοντέλα εφαρμογής. Πρώτον, διότι η απόδοση θέλουμε να διαχωριστεί και χωροθετικά. Δηλαδή, τι εννοώ, αν δει κανεί ότι ο κανονισμός αυτός ε, έχει εναρμονιστεί σε όλα τα κρατημέλη και ισχύει σε αυτά, απλά ισχύει παντού. Και το δεύτερο πλευρά ε, ουσία ε, είναι πιο σημαντικό και το υπογραμμίζει η κυρία Βέντεχο στην έκθεσή του. Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην απόδοση λόγω αμφισβήτησης και στην απόδοση λόγω ε, καταγγελίας της σύμβασης. Ο αγοραστής μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε δύο εβδομάδες, έχει την ε, δυνατότητα να παραιτηθεί ε, του προϊόντος χωρίς να έχει και το προϊόν ελάττωμα. Μετά από δύο εβδομάδες μπορεί να το πράξει αυτό, διότι απλά έτσι το επιλέγει. Όμως Όσον αφορά την ε, αμφισβήτηση, στις περισσότερες περιπτώσεις ε, αυτό αφορά τον πολιτή, τον πολιτή τον ίδιο. Σήμερα δεν έχω το χρόνο για να σε εξηγήσω τις διαφορές. Δεύτερο θέμα και θέλω και αυτό να το αναφέρω. Γιατί στο κεφάλαιο υπαριθμών 17 περιοριστήκαμε σε ένα ευσύνοπτο, σε μια ευσύνοπτη διατύπωση. Διότι εδώ πρόκειται για ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αναφέρεται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό το οποίο κεφάλαιο είναι πολύ περίπλοκο και πολύ μακροσκελές. Εμείς λοιπόν στη δική μας την πρόταση για το κοινό δίκαιο πολίσεων θελήσαμε να περιοριστούμε μόνο στα θέματα εκείνα τα οποία είναι σημαντικά για την ε, απόδοση ε, λόγω των ε, δύο προηγούμενων περιπτώσεων που σας ανέφερα, της ακύρωσης και της καταγγελίας. Και τέλος, επιτρέψτε μου να φέρω ένα τελευταίο σημείο. Η κυρία ε, πολύ σωστά είπε ότι γενικότερα το δικαίωμα του εμπλουτισμού και το δικαίωμα, ε, το δίκαιο του εμπλουτισμού, με και το δίκαιο της απόδοση, βρίσκονται μπροστά σε ένα αντίλημα. Ή να είναι ευσύνοπτα και κατανοητά και εύληπτα ή από την άλλη να επιφέρουν δικαιοσύνη σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί κανονισμοί είναι μακροσκελείς και περίπλοκοι. Εμεί, λοιπόν προσπαθήσαμε να προσθέσουμε ε, δύο ρήτρε. Και αυτό σημαίνει ότι αφενός έχουμε τη δική μας την προσέγγιση να έχουμε όπως σας είπα ένα ευσύνοπτο και εύληπτο κανονισμό και από την άλλη πλευρά με τις ρήτρε που προσθέσαμε να επιτύχουμε την απόδοση δικαιοσύνης και σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ähm, ähm, äh, λοιπόν, θα ήθελα καταρχήν ε, να ευχαριστήσω όλους όσοι μίλησαν για τις ιδιαίτερα εμπεριστατωμένες απόψεις τους. Και επιτρέψτε μου να συνοψίσω. Ε, πράγματι ασκήθηκε κριτική. Εγώ και από τις ε, δύο εισηγήσει θα ήθελα να επιλέξω δύο θέματα και να εστιάσω την προσοχή μου σε αυτό. Στην κυρία Βέντεχος, επιμερισμός κινδύνων και θέλω να σας πω ότι τουλάχιστον όπως εγώ ερμηνεύω το δίκαιο δεν τα βρήκα και τόσο αρνητικά αυτά που είπε. Επιμερίζεται ο κίνδυνος ανάμεσα στον πολιτή και τον αγοραστή. Αυτός ο επιμερισμός ε, κατά την άποψή μου πάντα είναι λιγάκι αυθαίρετος. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σε τελική ανάλυση και οι δύο ανεξάρτητα από απώλεια ή ζημιά και οι δύο να μην βρεθούν σε πλεονεκτική ή μειονεκτική θέση το αποτέλεσμα μετράει. Τώρα πώς θα επιμεριστούν οι κίνδυνοι αυτό ίσως ε, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Πάω τώρα στην έκθεση του κυρίου Βάκα και θέλω εδώ να ε, σχολιάσω το εξής. Είπε ότι τη στιγμή που ε, κατατίθεται μήνυση, κυρίως όσον αφορά τις προθεσμίες παραγραφής, κατά πόσον θα πρέπει να ανανοηθούν ή όχι, γιατί υπάρχουν αυτά τα δύο σχετικά συστήματα. Εδώ θέλω να πω ότι κάθε ένας από εμάς γνωρίζει ή το ένα ή το άλλο σύστημα. Και δεν θα προχωρήσουμε αν τσακωνόμαστε για το ε, κατά πόσον ε, θα πρέπει να παρατείνονται ε, τα χρονικά διαστήματα παραγραφής ή όχι. Υπάρχουν όπως σας είπα διαφορετικές απόψεις από αυτού, αλλά κατά την άποψή μου σε τελική ανάλυση αυτή η συζήτηση δεν βοηθάει εντάξει, εγώ αν θέλετε ε, σταματήστε ε, την παραγραφή ή ορίστε την εκεί που ισχύει ή ανανεώστε την. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Αυτά τα οποία μας είπατε σήμερα σε τελική ανάλυση είναι η προσωπική σας, η επιστημονική σας άποψη ή αυτά που μας είπατε στηρίζονται από το σύνολο των καθηγητών στο πανεπιστήμιό σας ή στη χώρα σας. Είναι προσωπική σας η άποψη ή όπως σας είπα την συμμερίζονται οι καθηγητές. Και αν ναι, ποιοι. εκφράζουν σήμερα την άποψή τους εδώ. Κατά τα άλλα θέλω επίσης να πω ότι οφείλει να είναι σαφές το πώς θα προχωρήσουμε. Εγώ έχω κάνει την εξής εμπειρία. Οποτεδήποτε ε, κάνει κανείς ερωτήσεις ε, σε καθηγητές πάντα ασκείται κριτική ο κάθε καθηγητής είναι σε θέση να συντάξει εκατοντάδες σελίδων για ένα αμεληταίο νομικό πρόβλημα. Μήνες μπορεί να συζητάει γι' αυτό. Στη Γερμανία τουλάχιστον αυτό ισχύει. Δεν ξέρω αλλού, αλλά εμείς στη Γερμανία ξέρετε έχουμε την τάση αυτή να το κάνουμε. Εάν λοιπόν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, είναι σαφές ότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αν δηλαδή αρχίσουμε σε κάθε μεμονωμένο άρθρο να μπαίνουμε στην ανθιποτελευταία ε, λεπτομέρεια, δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό. Και με τρόμο βλέπω την πλημμυρίδα των ε, τροπολογιών που θα υπάρξει, διότι ο κάθε συνάδελφος ε, θα αναφέρεται σε καθηγητές στη δική του την πατρίδα, θα αρχίσει να καταθέτει τροπολογίες, θα μας βομβαρδίσουν όλοι με τροπολογίες κατόπιν τούτου θεωρώ ότι πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε μια γραμμή. Είτε δηλαδή να τα θέσουμε σε ισχύ και τα, προγράμματα, τα προβλήματα ερμηνείας που ε, θα προκύψουν να τα παραπέμψουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή να δείξουμε εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα άρει τα προβλήματα που θα προκύψουν αν δεν σας αρέσει αυτό, να υπάρξει μια διακυβερνητική και εκεί να συμμετάσχουν οι καθηγητές πανεπιστημίου από όλα τα κράτη-μέλη και να τα βρούνε. Και όχι να προσπαθεί ο καθένας να ασκεί μονόπλευρα κριτική. Δεν υπάρχει άλλη λύση αν συνεχίσουμε με ακροάση επί ακροάσεων, δεν θα οδηγήσει αυτό πουθενά. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Κοιτάξτε, αυτό είναι το τελευταίο ε, εργαστήρι ε, για αυτό το πακέτο. Μετά θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, θα ξεκινήσουμε τι συζητήσει με τα Εθνικά Κοινοβούλια και κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ε, στη τελική ανάλυση δεν θα αποφασίσουν οι καθηγητές, εμείς θα αποφασίσουμε τι θέλουμε. Εκείνοι μπορούν να κάνουν εισηγήσει, αλλά εμεί θα αποφασίσουμε. Και έχω και μία ερώτηση σε αυτά που είπα είπαν Δηλαδή, αν ε, αυτή η απόλυτη προθεσμία παραγραφής των 10 ετών αφορά μόνο σπάνιες, ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, αλλά έχει προκαλέσει όλο αυτό το πολιτικό θόρυβο, ε, τότε γιατί δεν περιορίζεται το χρονικό διάστημα σε τέσσερα χρόνια. Να υπάρξει περιορισμός σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα παραγραφής, γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως σας είπα, πρόκειται για εξωτικές, όπως τις χαρακτηρίζει ο πρόεδρος, περιπτώσεις, ιδιαίτερα σπάνιες δηλαδή, τι έτσι κάνουμε αυτές. Να είναι πιο σύντομο το χρονικό διάστημα. Νομίζω εδώ μπορούμε να είμαστε πολύ σαφείς. Η κυρία Βέντεχορστ και μετά ο επόμενος ομιλητής. Ε, Φοβάμαι ότι θα πρέπει να σας απογοητεύσω, συνάδελφε. Αυτά που σας είπα εγώ δεν ήταν ε, άποψη καθηγητών, γιατί αν είχα εδώ να παρουσιάσω ακαδημαϊκή διατριβή, θα την παρουσίαζα τελείως διαφορετικά. Αυτά που σας είπα ήταν το απάβγασμα συζητήσεων με πολλούς νομομαθείς ε, που ασχολούνται με το θέμα αυτό αυτό είναι εξάλλου δικό μου συμπέρασμα. Και εγώ προσωπικά συμμετέχω σε ομάδα εργασίας για το Ευρωπαϊκό ε, Δίκαιο Πολίσεων και εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα και να πω ε, ότι το τι θα γίνει με τους κανονισμούς ένα και το αυτό. Σε τελική ανάλυση δεν παίζει ρόλο γιατί ένα πράγμα θα εφαρμοστεί. Κοιτάξτε, αν δεν καταστεί δυνατόν με αυτούς τους κανονισμούς να ρυθμίσουμε απλές ε, ε καθημερινές περιπτώσεις όπου παραδείγματο χάρη κατεβάζω μουσική από το διαδίκτυο, αν δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό ή κάτι άλλο πιο απλό, αγοράζω ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο που μου το παραδίδουν, ε, το συνδέουν και το πλυντήριο είναι ελαττωματικό. Αν λοιπόν αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε εμείς να τις λύσουμε ικανοποιητικά, τότε φοβάμαι ότι εδώ δεν πρόκειται για καθαρά ακαδημαϊκό πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Very, very... Πολύ σύντομα. θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι έχουμε δύο περίοδους παραγραφής, δύο χρόνια, δέκα χρόνια, η μία είναι υποκειμενική, η άλλη είναι αντικειμενική. Αλλά όπως σας είπα δεν υπάρχει κανόνας long stop. Και το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων επιτρέπει στα συμβαλόμενα μέρη να επιμικίνουν την δεκάχρονη περίοδο παραγραφής. Οπότε, αν το ΣΕΣΕΛ, το Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων, αφορά τη διαθέτηση των πωλήσεων και στόχο έχει να ρυθμίσει αυτές τις πωλήσει και ο βασικός, ε, το βασικό σημείο εδώ είναι η μη συμμόρφωση, υπάρχει ένας ευκολότερος ε, ρόλος στην ε, οδηγία για τις πωλήσει που λέει ότι η παραγραφή λαμβάνει χώρα δύο χρόνια μετά την παράδοση του αγαθού. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε τι γίνεται αν μετά από 8 χρόνια ο πολιτής ανακαλύψει ότι από την αρχή το αυτοκίνητό του είχε ένα ελάττωμα. Γιατί τώρα 8 χρόνια. Οπότε τι θα ισχύσει, ποια παραγραφή θα ισχύσει εδώ, 8 συν 2 10 χρόνια είναι η ανώτατη περίοδος παραγραφής ή αν τα συμβαλόμενα μέρη τροποποιήσουν την περίοδο παραγραφής μπορούν να την παρατείνουν σε 30 χρόνια για παράδειγμα αυτή την προθεσμία. Στην πράξη το ζήτημα είναι σημαντικό όχι μόνο για τα πανεπιστήμια και τους καθηγητές, νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους πολίτες, για τους ενδιαφερόμενους και χρήζει διευκρίνησης. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ τους δύο εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να καλωσορίσω θερμά τον Υπουργό ε, Εμπορίου Βιομηχανίας ε, και ετηρισμού ο οποίος ε, είναι αρμόδιος και για θέματα τα οποία εξετάζουμε εμείς, ε, θέματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας και εταιρικού δικαίου. Εχθές είχαμε εδώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης ε, και τώρα πλέον και με εσά θα ακούσουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Ευρωβουλευτές, κύριε Αντιπρόεδρε και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Τζούρι, κυρίες και κύριοι, η σημερινή παρουσία μου στο Ευρωκοινοβούλιο και συγκεκριμένα ενώπιον της Επιτροπής Τζούρι δίνει συνέχεια στην καθιερωμένη πρακτική να ενημερώνεστε από την Προεδρία του Συμβουλίου για τις προτεραιότητες και δράσεις που αναλαμβάνει να προωθήσει κατά τη διάρκεια της εξάμεινης συνδύασης στα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εταιρικού δικαίου. Όμω, πολύ πέραν τη ανταπόκριση μου σε καθιερωμένε πρακτικέ, η εδώ παρουσία μου είναι δηλωτική πράξη του σεβασμού μου απέναντι στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει για να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοκρατικότερη, για να πλησιάσει περισσότερο και να φουγκράζεται καλύτερα του πολίτε τη. Άλλωστε, κεντρικό μήνυμα και βασική προσπάθεια της Κυπριακή Προεδρίας είναι για μια καλύτερη Ευρώπη πρώτα και κύρια για τους πολίτες της. Από την έναρξη ενισχύωση τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχουν διευρυθεί οι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω συνομοθέτη με το Συμβούλιο. Ως η Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνουμε την ετοιμότητα μα να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να προωθήσουμε με επιτυχία του φακέλου που θα διαχειριστούμε το δεύτερο εξάμεινο του 2012 στου τομεί τη αρμοδιότητας μα με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και το τωρικό δίκαιο. Στην αρχική μου παρέμβαση συνοπτικά θα σας παρουσιάσω τις βασικές μας πολιτικές και τα επιμέρους θέματα που θα διαχειριστούμε κατά τους επόμενους έξι μήνες όπως συμφωνήθηκα στο πλαίσιο του τρίου της Προεδρίας. Προτού όμως προχωρήσω με την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής όπως επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πολωνική και Δανική Προεδρία για όλες τις προσπάθειες και την πρόοδο που έχουν συντελεστεί στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και ειδικά στην επίτευξη συμφωνίας επί του πακέτου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το οποίο ως γνωστό συζητείται για τρεις δεκαετίες στην κοινότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το δίκαιο πνευματική ιδιοκτησία, η στρατηγική Ευρώπη 2020 αποδίδει μεγάλη σημασία στον εξυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της προστασίας τη πνευματική ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτόμα βιομηχανία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίδευξη της ενιαίας αγοράς της πνευματική Ιδιοκτησία. Προ αυτή την κατεύθυνση οι προηγούμενε του Τρίου Πολωνία και Δανία έχουν εργαστεί μαζί σα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευθύατηση των προτάσεων όσον αφορά πρώτον την τροποποίηση τη οδηγία 206-116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διάρκεια προστασία του δικαιώματο πνευματική ιδιοκτησία και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων. Δεύτερον, την ανάθεση στο γραφείο εναρμόδηση στο πλαίσιο τη εσωτερική αγορά εμπορικά σχέδια, εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα ε, καθηκόντω συναφών με την επιβολή τη εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανωμένη στη σύγκληση Ευρωπαϊκού Παρατηρητήου για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία με εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Και τρίτον, την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένε επιτροπέμενε χρήσει των ορφανών Άμεση προτεραιότητα τη Κυπριακή Προεδρία για του επόμενου μήνε είναι να αεροστικοποιηθεί ένα πολύ σημαντικό πακέτο για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, το πακέτο για τα διπλώματα τεχνίας. Θα εργαστούμε εντατικά έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα να συνυπογράψουν τη συμφωνία για τη δημιουργία του ενιαίου δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνία κατά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα το Οκτωβρίου. Όπω όλοι κατανοούμε βέβαια, η υπογραφή τη συμφωνία δεν μπορεί να καταστεί δυνατή εάν δεν οριστικοποιηθούν τα κείμενα των δύο σχετικών κανονισμών. Παρά την τεράστια πρόοδο που σημειώθηκε από του αρχιούς κρατών και κυβερνήσεων για την έδρα του ενιαίου δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνία, οι εισηγήσει σχετικά με τη διαγραφή των άρθρων 6 και 8 του κανονισμού για τη θέσπιση ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα τη δημιουργία ενιαίου καθεστώτο προστασία των ευρεσιτεχνιών έχουν προκαλέσει καθυστέρηση στην υιοθέτηση του πακέτου αυτού. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Συμβούλιο δεν έχει οριστικοποιήσει ακόμα τι εσωτερικέ του διαβουλεύσει σχετικά με τι υγιεί αυτέ. Έχουμε αποφασίσει, προτού προχωρήσουμε με τι εσωτερικέ μα διεργασίε, να δώσουμε το χρονικό περιθώριο που απαιτείται για να συζητήσουμε το θέμα μαζί σα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την αναβολή τη ψηφοφορία του φαγγέλου αυτού στην Ολομέλεια, δίνοντα έτσι χρόνο για τι αναγκαίε διαβουλεύσει μεταξύ των δυο συννομοθετικών σωμάτων. Είμαι βέβαιος, ωστόσο, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε πως οι ισορροπίες της λυμμένης συμφωνίας των αρχηγών κρατών μερών και κυβερνήσεων είναι πολύ λεπτές. Το άνοιγμα εκ νέου της συμφωνίας σε αυτό το στάδιο είναι μια πολύ ασυνήθιστη κίνηση και σίγουρα δεν πρέπει να θεωρείται ότι θα δημιουργήσει προηγουμένου. Όμως, αν είναι κάποιο θέμα για το οποίο αξίζει να υπάρξει μια μικρή απόκριση από τις διαδικαστικές συνήθειες μας, τότε σίγουρα είναι αυτό το θέμα, το οποίο ολοκληρώσαμε μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις που κράτησαν 30 σχεδόν χρόνια. Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στο ίδιο πνεύμα συνεργασία και από πλευρά Ευρωκοινοβουλίου, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό ο φάκελο το συντομότερο δυνατόν με επιτυχία. Με την υιοθέτηση του νομικού πλαισίου για την προστασία του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί εισάξιος ανταγωνιστής στη διεθνή αρένα της έρευνας και της τεχνολογίας. Στόχος της Προεδρίας μας είναι η λήψη των απαραίτητων μέτρων για να έχουμε την πρώτη αίτηση κατοχύρωσης του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας αρχές του 2014. Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ψηφιακή άλλη μορφή η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατίθενται στο κοινό και πώς αποζημιώνονται οι δικαιούχοι. Η θέσπιση οδηγία που να προβλέπει ενιαίους κανόνες για την εποπτεία της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου των, εταιρικών, των εταιριών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί πρωτεροίδα της Κυπριακής Προεδρίας προγραμματίζουμε να εξετάσουμε στο Συμβούλιο την ελόγω πρόταση, η οποία βάσει πρόσφατη ενημέρωση θα εκδοθεί από την Επιτροπή στι 11 Ιουλίου. Η πρόταση αυτή, μαζί με το θέμα των διπλωμάτων ευρωτεχνία, είναι ανάμεσα στι δράσει κλειδιά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ω τέτοια θα, έχει, θα είναι και η αντιμετώπιση τη στο Συμβούλιο, όπου έχουν προβλεφθεί πέντε συναντήσει τη σχετική ομάδα εργασία για το διάστημα Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη. Ο εξυγχρονισμό και η ομοιογένεια στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων περί των κοινοτικών εμπορικών σημάτων είναι ένα άλλο ζήτημα στο οποίο χρήζει άμεση αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο πρώτος κανονισμός για το κοινοτικό εμπορικό σήμα θεσπίστηκε το 1993, ενώ η πρώτη οδηγία για τα εμπορικά σήματα υιοθετήθηκε το 1989 και από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει πλούσια νομολογία κατά την ερμηνεία τους. Στη βάση αυτών των δεδομένων είναι αυταπόδειχτη η ανάγκη αναθεώρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Οι προτάσει της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τα κοινωτικά εμπορικά σύμμετα αναμένεται να υποβληθούν στο Συμβούλιο για συζήτηση εντός του ερχομένου Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε τις σημαντικές τις προτάσεις αυτές, καθώς ο εξυγχρονισμός των εθνικών γραφείων και των διαδικασιών που ακολουθούν θα ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικότερα την οικονομία. Επιπλέον, θα καταστήσει το νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει ακόμα πιο ασφαλές και αποτελεσματικό. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το ζήτημα της ομοιομορφίας των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του πλαισίου των εργασιών των μόνιμων επιτροπών του Παγκοσμίου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο και υποχρέωση να κατευθύνει τις συζητήσεις για την παραγωγή καινούργιου δικαίου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας στα σωστά νομικά πλαίσια. Ιδιαίτερη έφαση θα δοθεί στις καινούργιες συνθήκες που τροχοδρομούνται αναφορικά με την προστασία των ραδιοτοπληροπτικών οργανισμών καθώς και με τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις για τα άτομα με προβλήματα όρασης ή τα άτομα με ειδικέ ανάγκες εκτύπωσης. Προς το σκοπό αυτό έχει προγραμματιστεί χρόνος εξέτασης των διαφόρων θεμάτων που χρήζουν συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σε ό,τι αφορά το εταιρικό δίκαιο. Το εταιρικό δίκαιο και η εταιρική διακυβέρνηση είναι η ακρογωνία λύθη για μια σύγχρονη και δυναμική οικονομία. Η συνεχής βελτίωση και εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση συμβάλλουν τα μέγιστα στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθιστώντας την επιχειρηματικότητα πιο βιώσιμη, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανταγωνιστούν με επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές, συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στην οικονομική ανάπτυξη. Το εταιρικό δίκαιο μεταξύ άλλων τομέων περιλαμβάνει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και του λογιστικού ελέγχου. Είναι συνεπώ απαραίτητο για την προώθηση τη ανάπτυξη και την ενίσχυση τη εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ενιαία αγορά. Η πρόταση για τη μεταρρύθμιση των λογιστικών οδηγιών αποσκοπεί στην απλούστευση, σαφήνεια και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων και στη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων έχει αναγνωριστεί ω μια από τι πιο επιβαρυντικέ κανονιστικέ υποχρεώσει για τι επιχειρήσει. Η μείωση των ρυθμιστικών και διοικητικών επιβαρύσεων μέσω τη απλοποίηση των λογιστικών κανόνων και των υποχρεώσεων χρηματοοικονομική πληροφόρηση κρίνεται επιβεβλημένη ιδίω για τι μικρέ επιχειρήσει. Παράλληλα, χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στι πληρωμέ που καταβάλουν οι εξοριστικές και δασικέ επιχειρήσει σε κυβερνήσει η εν λόγω πρόταση αποτελεί ένα από τους πυλώνες της πράξης για την ενιαία αγορά. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πρόταση οδηγίας για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και σχετικές εκθέσεις ορισμένων τύπων επιχειρήσεων, η οποία καταργεί και αντικαθιστά τις λογιστικές οδηγίες 78 του 660 και 83 349. Η πρόταση αυτή θα αποτελέσει προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία και θα εργαστούμε με στόχο την επίτευξη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε πως έχουν οριμάσει οι διεργασίε για να προχωρήσουμε στις μεταξύ μα διαπραγματεύσεις με προοπτική την υιοθέτηση της σε πρώτη ανάγνωση. Κατανοούμε και έχετε τη γενική στήριξη του Συμβουλίου στι ισχυρέ απόψει που εκφράζονται και εντό τη Επιτροπή αλλά και ευρύτερα εντό του Κοινοβουλίου για την εισαγωγή κανόνων διαφάνεια στι εργασίε των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στου τομεί των εξορίξεων και τη υλοτομία. Ταυτόχρονα όμω, η συνδεπτική πλειοψηφία των κρατών μελών είναι πεπισμένη πω θα πρέπει να εξεύρουμε μια συμβαστική φόρμουλα που θα κρατά τι ισορροπίε μεταξύ διαφάνεια και ανταγωνιστικότητα. Προσβλέπουμε στην επικοδημητική μα συνεργασία με τον Πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή και εισηγητή των κύριο Λένε, καθώς και τους κοιόδης εισηγητές, αλλά και σας των μελών, έτσι που στο τέλος να φτάσουμε στη συμφωνία σε πρώτη αγράμμιση. Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την πρόθεση των προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του λογιστικού ελέγχου που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τους υποχρεωτικούς λογιστικούς ελέγχους, στη βελτίωση της ποιότητας ε, του ελέγχου που διενεργείται και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτή άλλωστε είναι μια αναγκαιότητα που έχει αναδείξει η πρόσφατη οικονομική κρίση. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την έκδοση του σχεδίου έκθεσης κοινοβουλευτική σας επιτροπή περί τα μέσα Σεπτεμβρίου και προσλέπουμε στη στενή συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδη εισηγητές για πρόοδο στο σημαντικό αυτό φάκελο. Τέλο, Όσον αφορά στην πρόταση για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο, συμφωνώ με την άποψη ότι τα Ιδρύματα επιτελούν πολύτιμο έργο προ όφελο των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο αυτό πρέπει να εθαρρυνθεί και τα Ιδρύματα να βοηθηθούν να προσελκύσουν περισσότερη χρηματοδότηση. Η πρόταση του κανονισμού του Συμβουλίου για το θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο αποσκοπεί στη δημιουργία μια ενιαία ευρωπαϊκή νομική μορφή. Στόχος της είναι η διευκόλυνση της σύστασης των Ιδρυμάτων και η διασυνοριακή άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Η Κυπριακή Προεδρία, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή σας, θα εργαστούμε σκληρά για να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή πρόοδο σε αυτόν τον πολύ δύσκολο φάκελο. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς και την Επιτροπή για τη συμβολή σας το μπορεί να ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση και η συμφωνία σε ό,τι αφορά τα αφανά έργα και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεση σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Πράγματι αναφέρατε πάρα πολλά θέματα. Ε, έχουμε πλησιάσει σε πάρα πολλά εξ αυτών. Είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία. Υπάρχουν βέβαια κάποια εξ αυτών τα οποία είναι δυσκολότερα. Είναι δυσκολότερα και απαιτούν ε, πιο περίπλοκες διαπραγματεύσεις. Ζητήστε το το λόγο η συνάδελφη Κάριμ και ο συνάδελφος Μάση. Παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να καλωσορίσω τον Υπουργό στην Επιτροπή μας σήμερα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ε, έκανε τον κόπο τόσο νωρί να έρθει να συναντηθεί μαζί μα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κυπριακή Προεδρία, διότι έχει ήδη αποστείλει εκπροσώπου τη να συναντηθούν ε, και με μένα αλλά και με κάποιου άλλου συναδέλφου. Εμείς ως ε, Επιτροπή θα έρθουμε στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη εβδομάδα κύριε Πρόεδρο και προσβλέπω με ανυπομονησία στις ανταλλαγές που θα κάνουμε εκεί. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία τα οποία αναφέρετε στην ε, ε, παρέμβασή σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι μας δώσετε αρκετές πληροφορίες στην παρέμβασή σας. Επειδή υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι αναπάντεχα ευθύνη της ε, ε, Κυπριακής Προεδρίας. Πώς βλέπετε την πρόοδο του φακέλου για τους ελέγχους. Ε, πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να καταλήξετε σε συμφωνία πριν το τέλος της Προεδρίας σας. Και δεύτερον κύριε Πρόεδρε, αργότερα στη διάρκεια της ημέρας θα ψηφίσουμε την έκθεσή μου για την καλύτερη νομοθεσία. Και Λίγο πιο μετά θα γίνει και μια παρουσίαση της πρώτης αξιολόγησης αντικτύπου στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για ε, την ε, οδηγία που είχαμε για την αξιολόγηση αντικτύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα αναλάβετε κάποια βήματα ώστε να υπάρχει ένας αντίστοιχος μηχανισμός αξιολόγησης στο Συμβούλιο βάσει και της διαθεσμικής συμφωνίας. Κύριε Υπουργέ, τέλος, ακούσαμε και μία παρουσίαση ε, για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων προηγουμένω. Μάλλον είναι αυτό περισσότερο ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Αλλά επειδή έχετε κι εσεί κάποιο δρόμο, ρόλο να διαδραματίσετε για το εμπόριο, πώ ε, βλέπετε τη σχετική πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει το λόγο. Ε, ο επόμενο ομιλητή. Ο κύριο Μασιπιντάλγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Κυπριακή Προεδρία, διότι έκανε τον κόπο να έρθει μέχρι εδώ. Ίσως το γνωρίζετε, εγώ είμαι υποστηρικτής, ε, πολύ στεναρός υποστηρικτής των διεκδικήσεων της Κύπρου για τα κατεχόμενα και επομένω νιώθω ότι είμαι φίλος σας και γνωρίζω τη χώρα σας, γνωρίζω τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και θεωρώ ότι η Προεδρία σας θα είναι λαμπρή. Και από πλευρά μου να περιμένετε τη μέγιστη δυνατή συνεργασία. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε τόσο στη σημασία του πνευματικού δικαίου και στη σημασία των εμπορικών σημάτων ε, για το θέμα το οποίο έθιξε τώρα ο συνάδελφος Καρίμ για τις επιτροπές αξιολόγησης ε, και την αξιολόγηση αντικτύπου νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε ε, θα το συζητήσουμε και αργότερα εδώ στην Επιτροπή μας σήμερα το απόγευμα δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτό θα ήθελα όμως να σας πω το εξής Αναφερθήκατε στην καλή πορεία των εργασιών για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ε, και το τι έκαναν οι προηγούμενες προεδρίες. Με όλο το σεβασμό, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Νομίζω ότι το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ε, βρίσκεται ε, πλέον στα όρια της κατάρρευσης. Υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις σε κυβερνητικό επίπεδο και για μένα δεν αποτελούν καμία ικανοποίηση και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ε, αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα και νομίζω ότι ε, οι κυβερνήσεις ε, τραβούν στα άκρα το θέμα αυτό και φαντάζομαι ότι υπήρχαν εκπρόσωποι σα και στο τελευταίο, στην τελευταία συνεδρίαση της Κορεπόερ Ξέρετε ότι το θέμα έχει παγώσει και δεν ξέρουμε προς τα που οδεύουμε. Αυτό το θέμα των διπλωμάτων ε, ε, ευρεσιτεχνίας, εάν όντως ε, οι προηγούμενες προεδρίες, αντίθετα με τα όσα μας είπατε, είχαν κάνει κάτι και το είχαν αναλάβει η Προεδρία και το Συμβούλιο, πραγματικά θα είχαμε επιτύχει ίσως κάτι περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν κύριε Υπουργέ, επειδή η Κύπρος είναι μια χώρα στην οποία διαπίστωσα η δίσόμαση, ότι μιλάτε εξαιρετικά την αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιείτε η αγγλική γλώσσα ως προτεραιότητα θα έπρεπε ίσως να εξεταστεί η δυνατότητα να ενωθούν όλες οι χώρες και να μην λάβουμε υπόψη για παράδειγμα τους Ισπανούς επί τη βάση του μόνο την αγγλική γλώσσα. Ίσως να είναι μια δυνατότητα να έχουμε πιο αίσιο και να έχουμε μια οδηγία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, και μια ενιαία θέση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας διότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είμαστε στα όρια της κατάρρευσης λόγω της καταστροφής που έχουν προκαλέσει τρεις κυβερνήσεις. Τίποτα άλλο. Ο κύριος Βιέφκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την επίσκεψη σας σήμερα και για την παρουσίαση που μας κάνατε των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτά που μας είπε ο κύριος Μασίπ για τα διπλώματα βρυσιτεχνίας. Ο συνάδελφος παρουσίασε τη δική του γνώμη. Θα ήθελα να ακούσω όμως τη δική σας γνώμη και τη δική σας απάντηση. Τι συνέβη στην πραγματικότητα. Γιατί πραγματικά ανησυχούμε τα μάλα. Τόσα χρόνια δουλειά και κόπων, τόσες προσπάθειες που έγιναν και από τις προηγούμενες προεδρίες αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο κόπο κάναμε για να καταλήξουμε σε μια ορθολογική συμφωνία και συνεννόηση και ξαφνικά, ευνηδιαστικά, την τελευταία στιγμή και μάλιστα τη στιγμή που περιμέναμε να διευθετηθεί μόνο το θέμα της έδρας του δικαστηρίου των Δηλωμάτων ευρυσιτεχνίας ξαφνικά το Συμβούλιο λαμβάνει μια απόφαση που σφετερίζεται τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λα, λαμβάνει μια υπόθεση που θέτει υποερωτηματικό την καλή βούληση ε, του Συμβουλίου για ανέβρεση λύσης. Τι συνέβη δηλαδή στο Συμβούλιο μπορείτε να μας πείτε. Κατά τη γνώμη σας ε, όλοι όσοι ψήφισαν κατάλαβαν τη, την έννοια αυτών των αλλαγών. Γιατί πραγματικά αυτές οι αλλαγές που προτείνει το Συμβούλιο ουσιαστικά ανατρέπουν όλο το πακέτο των διπλωμάτων επιστεχνίας. Θα πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό. Ήξεραν τι ψήφισμα, τι ψήφισμα στο Συμβούλιο. Θα ήθελα πραγματικά να μας διαβιβάσετε τη γνώμη σας κύριε Υπουργέ. Θα ήμασταν άπειρα ευγνώμονες γι' αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά το θέμα των διπλωμάτων ευρυστιχνίας, να πω και εγώ κάτι. Ε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτά που είπαμε πέρυσι στην Τρόικα, στο Τρίο, τα άρθρα 6 και 8, εμένα δεν με διέφεραν καθόλου. Απλά και μόνο ε, διότι επαναλαμβάνονται. Όμως τότε οι νομικές υπηρεσίες ε, είπαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της ε, τριμερούς ότι για να εφαρμοστούν ε, τα άρθρα, ή διατάξει του 118 θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις επί της ουσίας του διπλώματων, των διπλωμάτων ευρυστεχνίας. Και για να συμβαστούμε είπαμε εντάξει να πάρουμε τα άρθρα 6 με 8. Επαναλαμβάνω όμως, εμένα καθόλου δεν με ενδιαφέρουν. Είτε περιλαμβάνονται είτε όχι, Όσον αφορά στο θέμα κατά πόσον τα χρειαζόμαστε για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αυτό είναι αδιάφορο. Όμως δεν είναι αδιάφορο το να διατηρηθεί ο κανόνας και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί εάν το, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 30 ολόκληρα χρόνια στο τέλος θέλει να γελιοποιηθεί, να, κάνει αυτό που δεν θα έπρεπε να κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή αποφασίζει για ένα πακέτο και τελικά επειδή δεν υπάρχει η απαραίτητη νομική βάση το πακέτο αυτό ορίζεται και αναφέρεται ως αβάσιμο, νομικά αβάσιμο. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή που προέκυψε. η αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σε αντίθεση με τις αρμοδιότητες που τους έχουν εκχωρηθεί αποφασίζουν κάποια στιγμή τα μεσάνυχτα να νομοθετήσουν. Κάνοντας κάτι τέτοιο ειδού τα αποτελέσματα. Άλλο είναι λοιπόν να κάθε κανείς τα μεσάνυχτα να ε, προσπαθεί ε, πάση θυσία να καταλήξει σε μια απόφαση έστω και καταφεύγοντας το γόρδιο δεσμό, άλλο αυτό και το να εξετάζει κανείς τα θέματα σοβαρά. Τραγική λοιπόν η κατάσταση. Ε, πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά στο εξής πρόβλημα. Είτε ε, τα άρθρα 6 έως 8 θα τα συμπεριλάβουμε ή έστω κάποια ε, στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το περιεχόμενο του ε, δικαίου αυτού, βέβαια εδώ εμπλέκεται και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ή αυτή είναι μια λύση. Ή υπάρχει και άλλη λύση, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Και εγώ δεν ξέρω πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Ίσως το καλύτερο είναι να πάμε καταρχήν διακοπές, να τα συζητήσουμε, να αφήσουμε τους εμπειρογνώμονες μας κατά τη διάρκεια του καλοκαίρι να σκεφτούν, ελπίζοντας ότι όταν θα επανέλθουμε όλοι το Σεπτέμβρη θα έχει ε, προκύψει ε, κάποια ε, καλή ιδέα. Αλλά πραγματικά όλοι ανησυχούν όσον αφορά αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά πρέπει να εξευρεθεί μια λύση. Σε τελική ανάλυση θα είμαστε επικοδομητικοί, αλλά όχι προσφέροντας το τίμημα της αξιοπιστίας μας και το τίμημα ότι όλο αυτό το πράγμα ενδέχεται να καταπέσει ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, λυπάμαι, ε, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω τη συζήτηση από την αρχή, ε, διότι παράλληλα συνεδριάζει η Επιτροπή Μεταφορών και έπρεπε εκεί να παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μου. Όμως, όπως ε, τα παρουσιάζετε εσείς, η κατάσταση ε, σε αυτόν τον τομέα είναι το λιγότερο θα έλεγα η λαροτραγική. Τι γίνεται δηλαδή. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αλλά μόνο κατόνομα. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή ένα τέτοιο δίπλωμα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. Απαράδεικτο αυτό, απαράδεικτο. Κάτι τέτοιο υπονομεύει το νόημα του κανονισμού. Εγώ λοιπόν ε, θεωρώ ότι εδώ δεν υπάρχουν και πάρα πολλές δυνατότητες. Εάν επιμείνει το Συμβούλιο σε αυτή τη διατύπωση, και αυτό θα το κάνει ίσως ε, λόγω των ισορροπιών στο Συμβούλιο. Εάν το κάνει αυτό το Συμβούλιο βλέπω τα πράγματα πολύ μαύρα και δεν βλέπω και φως στο τέλος του τούνελ. Οι κυβερνήσεις ε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά τοποθετήθηκαν, τοποθετήθηκα και εγώ όμως και άσκησα κριτική, διότι εμένα με ενδιαφέρει ένα πραγματικό, ουσιαστικό ευρωπαϊκό, κοινοτικό αν θέλετε, δίπλωμα ευρυστεχνίας που να του αξίζει το όνομα που θα φέρει. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να πούμε με απόλυτη σαφήνεια ότι αυτά που αυτή τη στιγμή κάνει το Συμβούλιο κατά την άποψή μου είναι αδιανόητα όλα αυτά είναι παντελώς αντιπαραγωγικά ως προς την τελική μας υπόθεση. Ελπίζω βέβαια ότι η σοφία του ε, Συμβουλίου ε, θα αποδείξει ότι αυτά που λέω δεν ισχύουν αλλά ξέρετε κάτι, ε, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει έξοδος από το δίλημα ούτε στο Συμβούλιο. Περιμένω μεγάλη αγωνία ότι θα συμβεί αλλά σας προειδοποιώ να μην δεχθούμε ημίμετρα μία μισή λύση, να μην θελήσουμε παστησία το συμβασμό, διότι ένα ε, κοινό ευρωπαϊκό ε, πακέτο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα είναι ουσιαστικό μόνο εφόσον έχει και σαφείς κανόνες. Διότι ό,τι προκαλεί νομική ανασφάλεια, ό,τι οδηγεί σε νομικά αμφίσιμες καταστάσεις οτιδήποτε λοιπόν παρεμφερές δεν είναι το σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω και ένα, ε, μια, ένα αυστριακό ρητό που λέει ότι οι συμβιβασμοί δεν μπορούν να σταθούν πάντα. Άρα δηλαδή τι σημαίνει αυτό ένα ημίμετρο, ένας μισοσυμβιβασμός μακροπρόθεσμα ε, θα στραφεί κατά του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές και να μην επιτρέψουμε ε, να προκύψουν άλλες ε, εξελίξεις. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν ένας οργανισμός να ε, χορηγεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, και μετά να τα ελέγχει και όλα αυτά να μην ισχύουν. Ε, στη δημοκρατία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ισχύει η κατανομή των εξουσιών και υπάρχουν ε, ελεγκτικά όργανα που δεν είναι απαραίτητα τα ίδια όπως εκείνα που λαμβάνουν τις ε, αποφάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Ε, δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτές τις εξελίξεις που διαφαίνονται διότι θα δυσχεράνουν περαιτέρω την κατάσταση. Και επιτρέψτε μου και κάτι άλλο. Θα αναφερθώ σε αυτή την ε, κατανομή των τριών υπομονάδων, δεν ξέρω πώς αναφέρονται αυτά, υπάρχει μια τέτοια πρόθεση. Ε, στην αρχή ε, πολλοί είπαν, μα κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα. Όλα αυτά δεν πρέπει να οδηγήσουν σε μια σύγχυση. Παρ' όλα αυτά όμως αποφασίζονται αυτές οι τρεις υπομονάδες, ο μιλήτρια, υπομονάδες λοιπόν, όπου σε τελική ανάλυση μπορεί να συμβεί το εξής Εκεί όπου τα πράγματα είναι απλά, εκεί τα πράγματα είναι απλά, σε μια αλφα χώρα να ισχύουν αλφα διατάξεις περί διπλωμάτων ευρυστεχνίας. Σε μια β χώρα όμως άλλες πάλι διατάξεις. Β διατάξεις. Όσον αφορά αυτή τη διαδικασία που προάγει το Συμβούλιο, εγώ ε, είμαι κάθετα αντίθετη κάθετα αντίθετη και την ευθύνη είναι σαφές, την φέρει αποκλειστικά και μόνο το Συμβούλιο και όχι εμείς. Σας ευχαριστώ. Κύριο Υπουργό, παρακαλώ. Συγγνώμη, συγχωρείτε, κύριε Βίξτρομ και μετά ο κύριος Υπουργό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ όλοι αναφέρονται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας και είναι και λογικό, διότι είναι το πρόβλημα που μας απασχολεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Θέλουμε να πάμε λίγο πιο πίσω για να δημιουργήσουμε το μέλλον. Θέλουμε να ανατρέξουμε στην ιστορία για να σκεφτούμε τι είναι αυτό το οποίο μας καθιστά ένωση. Μια άνωση ε, ανθρώπων που τους ενώνουν κοινέ αξίες. Και δεν είναι οι χώρες αυτές που πρέπει να ενωθούν, είναι οι κάτοικοί τους. Εμείς λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το κικαιώνα επιλέξαμε ένα δρόμο αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν το τίμημα και δεν θέλουν να αποφασίσουν που θα πρέπει να εδρεύει το δικαστήριο. Εμείς λοιπόν πρέπει να δεχτούμε μεν την κατάσταση, αλλά τα πράγματα δεν είναι ιδανικά για την Ευρώπη. Και ξέρουμε και πόσο μας επικρίνουν, διότι το Κοινοβούλιο έχει δύο έδρες και μεταφέρεται μεταξύ ε, Γαλλίας και ε, Βρυξελών. Και τώρα έχουμε ένα κοινοτικό δικαστήριο το οποίο θα είναι ε, σε τρία διαφορετικά σημεία. Προσέξτε όμως, πρέπει να σκεφτούμε λίγο λογικά. καταφέραμε ε, μετά από πολλές προσπάθειες να προχωρήσουμε μια πρόταση που για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, για τους δημιουργούς ε, είναι πολύ σημαντική. Είναι μια πρόταση την οποία την περιμένουν όλοι εδώ και δεκαετίες. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε τους εκνευρισμούς και τις απογοητεύσεις μας και να δεχτούμε το γεγονός ότι καταφέραμε να διανύσουμε όλη αυτή τη μακρά πορεία εδώ στο Κοινοβούλιο μπορούμε να είμαστε περήφανοι, διότι σε τέσσερις μήνες καταφέραμε να προχωρήσουμε τρεις εκθέσεις ε, με πολύ μεγάλη ε, συνένεση στην ψηφοφορία. Τώρα, το γεγονός ότι το Συμβούλιο συμπεριφέρεται διαφορετικά ε, χωράει πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει κρίση, για παράδειγμα ε, μια συζήτηση η οποία θα έπρεπε να γίνει και δεν έγινε ε, κάποιες ελλείψεις. Παρά όμως ε, τα αίτια ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι όλα αυτά αποτελούν εφαλτήριο για μια νέα συζήτηση και θα πρέπει να συζητηθεί από εκεί και πέρα διεξαδικά το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να δούμε όλες τις λεπτομέρειες μία προς μία. Θα ήθελα όμως να ε, ζητήσω από το Συμβούλιο να διατηρήσει αυτή την προοπτική, δηλαδή την προοπτική της ΕΕ Ενωμένης Ευρώπης μέσα στην πολυπλοκότητά της. Να προσπαθήσουμε να πάμε πέρα από τις αντιφάσεις και να ε, δείξουμε σθένος και πειθό και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης εκεί που ε, αυτή τη στιγμή κυριαρχεί η έλλειψη εμπιστοσύνης. Δεν μπορούμε να έχουμε ελλείψεις, ασάφεια και θεσμικά προβλήματα αυτής της μορφής. Πρέπει να προχωρήσουμε ε, με ισχυρή την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε εδώ γιατί υπηρετούμε έναν ευρωπαϊκό λαό που ζει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και αυτή είναι η δέσμευση η οποία θα πρέπει να κυριαρχήσει. Σας παρακαλώ λοιπόν να το σκεφτείτε όταν θα το συζητήσετε αυτό στο Συμβούλιο την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, θεωρώ ε, ήταν αναμενόμενο και φυσιολογικό η συζήτησή μας να επικεντρωθεί στα θέματα του διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και στο ενίο δικαστήριο ε, και γι' αυτόν θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές και τον κύριο Χιδάλκο και τον κύριο Τσιέφκα, την κυρία Λίχτεμπερκερ και την κυρία Γουίλστρομ για το ότι αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα. Όμως εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο, ο κύριος Λένε, ε, και είναι σημαντικό αυτό ότι είμαστε μπροστά σε μια ε, δύσκολη κατάσταση, αλλά μα δίνεται ευκαιρία να αφήσουμε λίγο χρόνο και τώρα με τι διακοπέ οι, οι νομικές υπηρεσίες να δουν αυτό το ζήτημα, να δουν ακριβώ πού μπορούμε να βρούμε μια συγκεκριμένη λύση. Ε, δεν είναι τυχαίο που είπα και στην εισαγωγή μου παρέμβαση είναι ότι ε, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο να γίνονται αποκλήσεις σε αυτή τη διαδικασία. Όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε μια δουλειά που έγινε όλο αυτόν τον καιρό ε, εκεί που υπάρχουν ακριβώς παρουσιάζονται κενά και αδυναμίες να αφήσουμε αυτή τη δουλειά να πάει χαμένη. Ε, θα πρέπει να κάνουμε απόκληση από τι συνήθεις μας διαδικασίες και να βρούμε λύση. Θα σας πω ότι ε, η Προεδρία του Συμβουλίου θα δουλέψει σε αυτή την κατεύθυνση μαζί σας ε, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την ίδια την Ευρώπη. Είναι το σημαντικό για όλους εμάς. Και εδώ θέλω να ε, σημειώσω ότι αυτό που είπε και η κυρία Σεσίλια ε, Γουίστρομ ότι ε, η προσπάθεια μας εμάς και ο Κύπρος επειδή αναφέρθηκε πρέπει να κρατήσουμε την ΕΕ Ευρώπη μέσα στην πολυπλοκότητα τη. Εμεί είμαστε μια μικρή χώρα ω προεδρεύουσα μπορεί και μπορούμε να είμαστε ένας αξιόπιστος διαμεσολαβητή. Και να σας πω ότι το μήνυμα μας για καλύτερη Ευρώπη καλύτερη Ευρώπη για του πολίτε της μπορεί να γίνει εφόσον θα έχουμε και περισσότερη Ευρώπη. Και περισσότερη Ευρώπη σημαίνει να μπορούμε να βρίσκουμε ε, συμβιβασμούς και εκεί που είναι δύσκολα τα πράγματα και εκεί που φαίνονται τα πράγματα πολύ ε, αξεπέραστα και ανυπέρβλητα. Όλοι κατανοούμε την ανάγκη να ε, λειτουργήσουν οι κανονισμοί και το ενιαίο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνία, Κατανοώ ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα αλλά θεωρώ ότι ε, μέσα από την ε, καλή βούληση και θέλω να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά το Ευρωκοινοβούλιο για την αβολή της συζήτησης και την αποφάση στην Ολομέλεια γιατί μας δίνει την δυνατότητα και τον χρόνο ε, όπως είπε και ο Πρόεδρος ο κ. Δένε να, βρούμε λύσεις. Ε, τώρα στα άλλα θέματα να πω σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος ε, για το θέμα της ε, ε αξιολόγησης αντιτύπου. Ε, θεωρώ ότι το θέμα της αξιολόγησης αντιτύπου είναι ε, ένα θέμα το οποίο η Κυπριακή Προεδρία υποστηρίζει τη βελτίωση της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών ελέγχων και την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης. Εμείς στοχεύουμε ε, να ε, θεωρούμε ότι οι δύο προτάσεις ε, συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται και θα προσπαθήσουμε να, μέσα από τη στενή και επικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παράλληλα πάντοτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρούμε λύσεις και να σας πω ότι οποιαδήποτε έγγραφα εκδοθούν από το Ευρωκοινοβούλιο θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην επεξεργασία ε, αυτών των ε, προτάσεων. Ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα των φακέλων για τους ελέγχους, είναι, θα έλεγα ότι είναι, εύκολο είναι δύσκολο να ολοκληρωθούν πριν το τέλος της Προεδρίας. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει και οι δύο και ο κανονισμός και η οδηγία πρέπει να λειτουργήσουν παράλληλα και θα προσπαθήσουμε, είναι πολύ σημαντικό και για τις επιχειρήσεις και για την Ευρώπη και θα προσπαθήσουμε στον δυνατόν να προωθήσουμε ε, αυτούς τους ε, φακέλους. Ε, Θεωρώ αυτές ήταν οι απαντήσεις και αν υπάρχουν άλλες ευρύσεις και πρόεδρε είμαι στη διάθεση να σας απαντήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε και άλλες ερωτήσεις. Από ό,τι φαίνεται όχι. Κατόπιν τούτου ευχαριστώ θερμά τον κύριο Υπουργό. Ε, σας εύχομαι σε εσά και στην Κυπριακή Προεδρία καλή επιτυχία και εμείς από πλευράς μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλλουμε έτσι ώστε οι έξι μήνες να στεφτούν από επιτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Η ψηφοφορία τώρα είναι στις 11 ε, και δεν έχει τώρα νόημα να ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν διακόπτω τη συνεδρίαση μέχρι τις 11 και θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Μισό λεπτό. Ε, να πάρετε όλοι τις ε, κάρτες σας, γιατί όποιος δεν έχει την κάρτα του έχει περίπου 10 λεπτά να ε, βρει την κάρτα του.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 Παρακαλώ, κύριε και κύριοι, είναι 11 η ώρα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες μας. Θα ψηφίσουμε πρώτα την έκθεση του κυρίου Καρίμ. Έχετε κύριε Καρίμ κάποιες παρατηρήσεις για την έκθεσή σας μήπως? Ή μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Η γραμματεία με ενημερώνει ότι υπάρχει συνένεση. Δηλαδή, μπορούμε να ψηφίσουμε ομαδών τις τροπολογίες και το σύνολο της πρότασης του εισηγητού. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, οπότε ψηφίζουμε άπαξ τη γνωμοδότηση του κυρίου Καρίμ. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, δύο αποχές, Συγχαρητήρια κύριε Καρίμ. Επόμενο θέμα. Έκθεση του κυρίου Μεσάρος. Η γραμματεία δεν μου έχει δώσει συγκεκριμένε ε, πληροφορίες, οπότε θα ψηφίσουμε κάθε τροπολογία ξεχωριστά. Δεν θα καταμετρώ τις αποχές, ο συνήθως αλλά θα τις λάβουμε υπόψη στην τελική ψηφοφορία. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 12 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 6 υπέρ, κατά, 2 κατά, ε, εγκρίνεται. Πάμε στη 16 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 17 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 7 η συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 19 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 20 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 34 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 35 υπέρ κατά απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά ε, απορρίπτεται. Η 39 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για τη γνωμοδότηση στο σύνολό της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην άλλη έκθεση. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 14. Υπέρ, κατά, <laughs> πλειοψηφία Λοιπόν, οι δύο υπέρ, οι 15 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, οι 16 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 18 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 19 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 20 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 21 υπέρ κατά εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 3 η συμβαστική υπέρ, κατά, ένας κατά, εγκρίνεται. Η 24 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 8 υπέρ, κατά η 9 υπέρ κατά εγκρίνεται η τέσσερα συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται η 11 υπέρ κατά ε, εγκρίνεται, η 12 υπέρ κατά εγκρίνεται και αυτή. Τώρα ψηφίζουμε για τη γνωμοδότηση στο σύνολό της υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίθηκε ομόφωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια ε, στον εισηγητή. Πάμε στην έκθεση της Βιέφκα. Ψηφίζουμε. Εντάξει. Η 5 αποσύρθηκε. Έχουμε την 21. Υπέρ, κατά, αποχές. Ε, υπέρ, υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Η 24 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η συμβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 15 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 16 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 18 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 1 υπέρ, κατά, 19 δεν υπάρχει, είναι πιο κάτω. Γιατί την 1 τώρα, στο 1 είμαι. Υπέρ, Μισό λεπτό, στο ένα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Α, δίκιο είχατε. Ο συνάδελφος Ράπκα είχε δίκιο. Δεν έπρεπε να ψηφίσουμε για την ένα. Δίκιο είχατε. Άρα η ένα δεν έλαβε χώρα. Πάμε στη 19. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε στην 4 και αγνοούμε την 20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για τη γνωμοδότηση στο σύνολό τη, Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Πάει και αυτό. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάμε την αναφορά τα ορφανά έργα. Θέλετε να τοποθετηθείτε επ' αυτού, παρακαλώ. Η κυρία Γκέριγκερ Ντεόντεμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το πέρας των διαπραγματεύσεων στο Συμβουλίο με τη Δανική Προεδρία, ακόμη ήταν επί Δανικής Προεδρίας. Ε, τότε έγιναν οι συζητήσεις για ελεύθερη χρήση των ορφανών έργων στις 6 ε, Ιουνίου ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο και η συμβαστική λύση έγινε δεκτή στις 14 Ιουνίου στην Κορεπέρ. Εν συνεχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπλήρωσε την σχετική τεκμηρίωση και μας την έστειλε στις 20 Ιουνίου. Τώρα έχουμε συμπληρωμένο το πακέτο, ενωπημένο το έγγραφο, καλό κατά τη γνώμη μου καταφέραμε να καταλήξουμε σε πραγματικά δόκιμες συμβαστικές λύσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους και ηγητές για την αγαστή συνεργασία, την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Χάρη σε αυτήν καταφέραμε να καταλήξουμε σε καλό, σαφές και χρήσιμο κείμενο, όπως είναι το κείμενο της νέας οδηγίας που με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Για τελευταία φορά σήμερα έχουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για την ε, Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω σήμερα να υπερψηφίσουμε τη συμβαστική πρόταση. Επαναλαμβάνω, είμαι πεπισμένη ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η πρόταση και ε, ήρθα σε επαφή με τηλεοράσει, με αρχεία, με βιβλιοθήκε. Είναι πολύ ικανοποιημένοι με το κείμενο και στο μέλλον θα χρησιμοποιήσουν πολύ ευχαρίστω αυτή την οδηγία. Λοιπόν, προτείνω να υπερψηφίσουμε, επαναλαμβάνω το κείμενο. Ευχαριστώ. Λίχτενμπεργκ, παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι μάλλον απογοητευμένη από το αποτέλεσμα. Διότι σε τελική ανάλυση αυτά τα οποία περιμέναμε. Δηλαδή ε, να υπάρχει προσπελασιμότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και κάτω από ιδιαίτερες εθνικές ε, προϋποθέσεις. Με την, ε, προϋποθε... με την μεταρρύθμιση των IPR ε, αν αρχίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποφασίζουμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει, ό,τι θέλει δηλαδή, ε, και εδώ αναφέρομαι στα κράτη-μέλη, τότε δεν θα υπάρχουν πλέον ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Ξέρω ότι ήταν ε, δύσκολες οι διαπραγματεύσεις και ξέρω ότι η συγγήτρια προσπάθησε να διαφυλάξει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά θέλω να πω ότι αν το Συμβούλιο συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, τότε τους στόχους που έχουμε θέσει, παραδείγματο χάρη όσον αφορά την εναρμόνιση των εξαιρέσεων, δεν θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένη από τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο χειρίζεται το θέμα αυτό. Και αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι που είχαμε θέσει, ε, που δεν είδαν επιτεύχθησαν και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε την ειλικρίνεια να το δεχόμαστε αυτό. Ε, πρόεδρος, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε σήμερα επ' αυτού, ε, μόνο να επιληφθούμε του θέματος. Άρα λοιπόν επιληφθήκαμε του θέματος και θα ε, διαβιβάσουμε την απόφασή μας στην Ολομέλεια. Green παρακαλώ. Καταλαβαίνω σε κάποιο βαθμό την απογοήτευση των πρασίνων, της ομάδας των πρασίνων. Αλλά δεν συμφωνώ ότι είναι δύσκολη η νομοθεσία. Εγώ το αντίθετο. Πιστεύω ότι καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση στα ορφανά έργα που ήταν ε, τελείω μπλοκαρισμένη γιατί ήταν ε, ανύπαρκτη η πρόσβαση. Είναι η πρώτη χρονιά, είναι το πρώτο βήμα πολύ δύσκολο που κάναμε μετά από αυτές τις επίπορες διαπραγματεύσεις. Η συνέχεια θα είναι πολύ πιο εύκολη. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη από την άποψη αυτή και θεωρώ ότι θα πρέπει να δεχτούμε σήμερα το κείμενο προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα για να εφαρμοστεί στη συνέχεια και εμπράκτο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπερλίνγκουερ. Θα ήθελα κι εγώ να σας πω την άποψή μου. Διότι το έργο της συναδέλφου Λίδια μας οδήγησε σε αποτέλεσμα παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες στιγμές που θεωρήσαμε ότι δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Και αυτή είναι αξιολόγηση. Έχουμε αποτέλεσμα πλέον. Αυτό που θα περάσουμε στην Ολομέλεια σήμερα θα είναι αποτέλεσμα. Αν καταφέρουμε να έχουμε ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση και το Συμβούλιο δεν αλλάξει για άλλη μια φορά στάση όπως συνήθως ε, ε διαπιστώνουμε, το γεγονός ότι θα υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, ευρωπαϊκή οδηγία για τα ορφανά έργα αποτελεί καινοτομία. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ευρώπη τα μεγάλα βήματα δεν γίνονται ξαφνικά. Αυτά τα βήματα τα οποία δίνουν την εντύπωση ότι είναι ανεπαρκή αλλά τελικώς ε, οδηγούν σε θετική πρόοδο είναι αυτά τα οποία μας οδηγούν στην εξέλιξη. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να έχουμε, αν όχι σε όλες τις χώρες, στις πιο προηγμένες χώρες, μία μορφή ψηφιοποίηση των ορφανών έργων και μία δυνατότητα να τα εξετάσει κανεί ε, στο διαδίκτυο θα αποτελέσει μία πολύ σημαντική καινοτομία. Ούτε κι εμεί είμαστε ικανοποιημένοι στο 100%. Ε, κατανοώ απολύτω τι παρατηρήσει τη ΕΒΑ. Αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να μα ε, οδηγήσει στο να απορρίψουμε και τι θετικέ πτυχέ. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τη Λίβια για το έργο τη και για όλου όσου συνεισέφεραν σε αυτό. Και εγώ θέλω να υπογραμμίσω εκ μέρους των φιλελευθέρων ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν ιδιαίτερα επίπονες ε, και χρονοβόρες. Ε, ναι. Και στην αρχή ήταν και αρκετά περιορισμένες. Μετά όμως ε, συνεχίστηκαν έγιναν κουραστικές. Υπήρχαν και πάρα πολλές τριμερείς ε, συζητήσεις. Ε, νομίζω ότι για τα ορφανά έργα, εκτός από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εκεί είχαμε τις περισσότερες ε, διαπραγματεύσεις. Συμπεριλάβαμε και τα ΣΔΙΤ, έτσι ώστε και οι βιβλιοθήκες και τα Ινστιτούτα να έχουν τη δυνατότητα με βοήθεια από την ιδιωτική οικονομία να προχωρήσουν στο έργο ψηφιοποίησής τους. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι τόσο περίπλοκα. Ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εξαιρουμένων των ταινιών. Αυτά εκεί είναι πιο δύσκολα. Όσον αφορά όμως τα βιβλία, νομίζω ότι πράγματι όλα αυτά μπορούν να ψηφιοποιηθούν και η εισηγήτρια ε, πάρα πολύ καλά συνόψισε τις διάφορες θέσεις. Και εγώ θα ήθελα εκ μέρους του ΕΛΚ να εκφράσω την υποστήριξή μου προς την κυρία Γκέριγκερ. Γιατί έκανε ό,τι μπορούσε, δεν επίστη προσπαθειών για να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα μιας συμβαστικής λύσης και μια συμβαστική λύση εξορισμού δεν μπορεί να ικανοποιεί τους πάντες. Αλλά συμφωνώ ότι κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα και νομίζω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε την κυρία Γκέριγκερ. Ο κύριος Έγκστρομ, ο τελευταίος ομιλητής. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου από την οδηγία αυτή. Ε, συνεργάστηκα στενά με τις βιβλιοθήκες και δεν είναι καθόλου ικανοποιημένες ε, με την οδηγία. Θεωρούν την οδηγία άχρηστη ή σχεδόν άχρηστη. Βέβαια, αν υπάρχει ε, η ε, μεγάλη πλειοψηφία να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία από ό,τι φαίνεται θα υποκληθώ αλλά κρίμα δεν νομίζω να συμβάλλουμε στο να γίνει προσιτή η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά θα ήθελα να απευθύνω έκκληση να επανεξετάσουμε το θέμα μπορούμε να το περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση γιατί με τη μορφή που έχει τώρα η οδηγία δεν είναι καθόλου χρήσιμη δυστυχώς Πολύ ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Άρα επιληφθήκαμε του ε, θέματος. Ε, κατόπιν τούτου το όλο θέμα θα παραπεμφθεί στην Ολομέλεια και η Ολομέλεια θα έχει τον τελευταίο λόγο, όπως συμβαίνει πάντα. Πάει το 21 και πάμε τώρα σε αυτή την περίπτωση της επιστολής. Ε, δεν ξέρω αν έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την αναφορά αυτή. Από ό,τι βλέπω όχι. Μισό λεπτό. Ο συνάδελφος Σπυρώνη έχει το λόγο. Δεν έχω βασικές ενστάσεις ε, καταρχήν, αλλά δεν κατάφερα να βρω τίποτα στη δεκμήριασή μου. Πώς θα ψηφίσω, διότι εδώ μου λείπει το σημείο 22 στο φάκελο και δεν ξέρω γιατί μιλάμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια συγκεκριμένη επιστολή. Κανονικά πρέπει να έχει διανεμηθεί αυτή. Αν δεν έχει διανεμηθεί, παρακαλώ να το πράξετε και θα ψηφίσουμε αργότερα. Όχι, έχει διανεμητή η επιστολή. Με mail, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κύριε Σπυρώνη, αν θέλετε, θέλετε να το αφήσουμε κατά μέρο και να επανέλθουμε αργότερα, να ψηφίσουμε αργότερα. Τι θέλετε, να ψηφίσουμε και το απόγευμα, αν θέλετε. Μένα δεν με νοιάζει, λέει ο πρόεδρος. Α, το βρήκα ε, δεν ήταν στο φάκελο εκεί που το ψάχνα. Πολλέ φορές είναι δύσκολο, μπερδεύω τα έγγραφα και δεν μπόρεσα να το βρω. Κατόπιν ε, ζητώ συγγνώμη και αποσύρω την επιφύλαξή μου. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος, αλλά δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Αποφασίσαμε και από αυτού και πάμε τώρα στη νομική βάση. Και ξεκινάμε με πρόγραμμα δράση ε, θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνία και τη φορολογία κτλ. Συνάδελφε Φως, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτή την πρόταση κανονισμού πρόκειται για τα νέα δασμολογικά και φορολογικά προγράμματα για την περίοδο μέχρι το 2020. Τα δασμολογικά και τα φορολογικά ρυθμίζονται σε δύο διαφορετικές ξεχωριστές νομικές πράξεις. Αυτό το ήθελε και το Κοινοβούλιο και γι' αυτό το Μάιο η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να ε, θεσπίσει δύο διαφορετικές εκτέσεις. Τώρα το θέλει και το Συμβούλιο και έτσι λοιπόν η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να στείλει δύο διαφορετικές εκτάσεις. Το, η, η Επιτροπή ΙΜΚΟ ζήτησε εμάς, ρώτησε εμάς ε, πώς θα κατανεμηθούν αυτές οι προτάσεις. Η μέχρι τούδε απόφαση βασίζεται σε διπλή νομική βάση, δηλαδή στο άρθρο 33 και στο άρθρο 114. Το άρθρο 33 ασχολείται με τα μέτρα συνεργασίας στον τελειωνιακό τομέα και το 114 αφορά την εναρμόνιση των ε, διοικητικών διατάξεων για την λειτουργία της κοινή αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση αυτή αφορά δύο βασικούς στόχους, τα άρθρα 113 και 114 Είναι η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Τώρα, το ποιο θα είναι το κείμενο το τελικό, αυτό δεν το ξέρουμε, απλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα άρθρα 33 ε, και 114 θα είναι τα ίδια και για το κομμάτι το φορολογικό. Αυτή λοιπόν τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτά τα δύο άρθρα ε, να βασίζονται στην ισχύουσα διπλή νομική βάση. Επειδή όμως έχει ανακοινωθεί ε, ο διαχωρισμός ε, των προτάσεων, γίνεται επεξεργασία των κειμένων και γι' αυτό λοιπόν συστήνω στην Επιτροπή μας να δώσει την εξής απάντηση στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Στο βαθμό που χρειάζεται θα δοθεί απάντηση μόλις έχουν κατατεθεί και οι σχετικές προτάσεις. Νομίζω πολύ σοφή η πρότασή σας, λέει ο αναβολή λοιπόν. Άρα αναβολή και πάμε ε, στο δεύτερο ε, που είναι πάλι ο συνάδελφος ε, Φως πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο, στα άρθρα 42 και 43 της συνθήκης και η Γεωργική επιτοπή Επιτροπή ε, καλεί την Νομική Επιτροπή να διευκρινίσει την νομική βάση, δηλαδή άρθρο 42 και άρθρο 43 παράγραφος 2. Η καταλληλότητα της ε, νομικής ε, βάσης δεν αμφισβήτηται από εμάς, απλά πρόκειται για διευκρίνηση και το άρθρο 43 αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής ε, των κανόνων του ε, ανταγωνισμού. Το άρθρο 42 αφορά τη νομική βάση για μια κοινή γεωργική πολιτική, ε, κάτι το οποίο έχουμε κάνει επανειλημμένα. Τώρα, οι άλλες παράγραφοι του άρθρου 43 που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής, αυτά ρυθμίζουν άλλα θέματα. Κατόπιν τούτου εγώ προτείνω στην Επιτροπή τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 να επιβεβαιωθούν ως ε, ε, η κατάλληλη νομική βάση. Καμία αντίρρηση. Άρα αποφασίζεται και αυτό. Πάμε στο 38. Όχι, αναβλήθηκε και αυτό. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος. Πάμε στο 25. Πρόκειται για αναδιατύπωση του Ενωσιακού Τελωνιακού Κώδικα. Αναβλήθηκε μόνο η απόφαση, κύριε Λίχτεμπεργκερ, αλλά είναι εδώ η νομική υπηρεσία και θα μπορούσαμε ίσως να ακούσουμε την άποψη της νομικής υπηρεσία διότι αφορά την πολιτική αλληλείας και εξαιρέσει για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Υπάρχει ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και είναι ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε την επόμενη φορά, αλλά καλό θα ήταν οι παριστάμενοι να ακούσουν την ε, άποψη της νομικής υπηρεσίας, διότι είναι περίπλοκο το ζήτημα. Καλό θα ήταν λοιπόν να ακούσουμε την ε, άποψή τους. Θα μπορούσαμε ίσως να τους δείσουμε να λάβει το λόγο. Εγώ ερωτώ, μπορεί αυτό να το κάνει σήμερα η νομική υπηρεσία ή να το κάνουμε την επόμενη φορά, στην επόμενη συνεδρίασή μας το Σεπτέμβριο. Ίσως και τη συζήτηση ολόκληρη θα μπορούσαμε την να βάλουμε για το Σεπτέμβριο. Αυτό είχαμε καταλάβει κι εμείς, ότι είχε αναβληθεί το θέμα. Okay, Πολύ ωραία. Ε, άρα, κυρία Λίχνιμπεργκ, επειδή δεν είναι έτοιμη, να το κάνουμε το Σεπτέμβριο. Δεν έχει νόημα αλλιώ. Πάμε στο 25. Πρόκειται για αναδιατύπωση. Ο συνάδελφος ε, Λόπε Ιστόρες. Παρακαλώ. Δεν έχει τίποτα να πει. Έχουν υποβληθεί όλα σε γραπτή μορφή. ένα πρόβλημα. Αν λοιπόν δεν έχετε αντιρρήσεις, θεωρώ ότι ελήφθη απόφαση. Έτσι κι αλλιώ, ε, αν δεν κάνω λάθο. Αναβάλαμε τις ε, κρατικές ε, προμήθειες τις δημόσιες συμβάσεις, ε, αναβολή της έκθεσης Μπαλντασάρ. Πάμε τώρα στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Και άκουσα ότι δεν έχει έρθει ακόμα το Συμβούλιο γιατί προβλεπόταν η συζήτηση για τις 12 παρατέταρτο. Ούτε ο κύριος Πενέρα είναι παρόν. Άρα δηλαδή ας περιμένουμε λιγάκι τον επικεφαλής της νομικής υπηρεσία και το Συμβούλιο και όταν θα έρθει το Συμβούλιο μπορούμε να ξεκινήσουμε έχετε κάτι άλλο, τα άλλα να τα συζητήσουμε καλύτερα σήμερα το απόγευμα. Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα για ένα τέταρτο. Μέχρι να έρθουν όλοι, κυρία Βίξτρομ. Μήπως θα έπρεπε να ψηφίσουμε και για την άρση της ασυλίας. Όχι. Ναι, αλλά αυτό και κλεισμένο το θηρών. Και έχουμε και την ακρόαση Colin Langen, αλλά αυτό τεχνικά δεν γίνεται. Δεν έχω τίποτα άλλο στην ημέση διάταξη που θα είχε νόημα να το εξετάσουμε τώρα. Τι να κάνω εγώ τώρα, λέει ο πρόεδρο. Θα μπορούσαμε το πολύ πολύ να εξετάσουμε το 35. Αλλά δεν ξέρω αν είναι παρόντες όλοι οι συζητητές. Πρόκειται για την έκθεση Lichtenberger. Αν θέλετε μπορούμε να εξετάσουμε αυτό το θέμα που δεν θα διαρκέσει και πολύ. Εντάξει κύριε Λίχτινμπέργκε θέλετε να το συζητήσουμε τώρα το θέμα σας. Και το 36 και αυτό στα γρήγορα μπορούμε να το εξετάσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βρήκαμε ένα θέμα μερίσια διάταξη για να ασχοληθούμε. Τα σπέσια, λέει ο πρόεδρος. Και η κυρία Λίχνιμπεργκα έχει το λόγο. Δεν θα θυμάμαι απ' έξω, λέει και η κυρία Λίχτινμπράγκα. Πρόκειται για αυτόν τον κανονισμό. Είναι μια γνωμοδότηση για περαιτέρω εξέταση και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι στον τομέα αυτό να ε, έχουμε κατά νου εξής. Ποια υλικά παίζουν ρόλο εδώ. Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όπως επίσης και το καθοριστική σημασία σε θέμα της αστικής ευθύνης. Αστική ευθύνη όταν υπάρξουν στην περίπτωση ύπαρξη ατυχημάτων με ε, βαριές Εγώ θέλησα να υπάρξουν διευκρινήσεις σε αυτά τα θέματα. Τροπολογία 2. Είναι πολύ σημαντική. Ευθύς εξ ε, να ερευνάτε το κατά πόσον κάποιος που λαμβάνει μία εντολή κατά πόσον ε, είναι φερέγγιος να μπορεί να αποζημιώσει στην περίπτωση που χρειαστεί. Δηλαδή είναι σημαντικό ευθύς εξ αρχής να γνωρίζουμε τις οικονομικές δυνατότητες του παραχωρησιούχου. Ε, θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να αναθέσουμε σε κάποιον ένα έργο ο οποίος όμως δεν είναι σε θέση ούτε να συνάψει ασφαλιστικά συμβόλαια ούτε να καταβάλει τα προσαποζημίωση ποσά οποτεδήποτε προκύψουν ζημιές που έχει ο ίδιος προκαλέσει. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι το εξής. Πρέπει σε όλον αυτόν τον τομέα να αναζητούμε τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Best available techniques λέει η ομιλήτρια, όχι technologies. Δηλαδή αυτό που έχουμε ε, διασφαλίσει ε, στα κράτη-μέλη Αυτά όλα πρέπει να κατοχυρωθούν έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούμε πεπαλαιωμένες τεχνολογίες οι οποίες έχουν αποδειχθεί ότι είναι, και, ε, ότι είναι επιβλαβείς, ότι προκαλούν βλάβες. Παναλαμβάνω λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι η φερεγγιότητα, η οικονομική επιφάνεια ε, των επιχειρήσεων και εγώ αυτό ε, θα το ξαναναφέρω στις τροπολογίες μου. Εμείς από ευρωπαϊκής ε, πλευράς επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι ιδιαίτερα όσον αφορά σε οικολογικά ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές είναι απαραίτητο να υπάρχει ιδέουσα προσοχή γιατί πρόκειται για την προστασία όχι μόνο του ε, θαλάσσιου αλλά και του παράκτιου πλούτου. Και οι ζημιές ε, δεν προκαλούνται μόνο για την αλία αλλά και για τον τουρισμό, κυρίως για τον τουρισμό, οι συνέπειες μπορεί να είναι τραγικές, ολέθριες. Εγώ λοιπόν αναφέρω αυτές, αυτές τις προστατευόμενες περιοχές ε, στο θαλάσσιο τομέα. Αναφέρομαι στην οδηγία περί ε, οικοτόπων, περί προστασίας ε, πτηνών, γιατί υπάρχει μία τάση είτε να αγνοείται παντελώς η νομοθεσία περί περιβάλλοντος ή αν λαμβάνεται υπόψη να προκαλούνται ζημιές όπου εκ των υστέρων κανείς δεν μπορεί να διαπιστώσει ποιος καλείται να αποζημιώσει. Αυτά είχα καταρχήν να πω και όπως ε, σας είπα το σημαντικότερο εξ όλων είναι να επισημάνουμε ότι υπάρχει ε, ανάγκη προστασίας, ε, είναι απαραίτητο ε, κάποιος να αναλαμβάνει την οικονομική ευθύνη και αυτό να καθίσετε σαφές ευθύς εξ αρχής έτσι ώστε να μην εκ των υστέων, να μην καλείται κανείς να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες καταστάσεις. Στον τομέα αυτό υπήρξαν πάρα πολλά ατυχήματα, γνωστές είναι οι ζημιές που έχουν προκληθεί και όπου ορισμένες χώρες που επλήγησαν κυρίως οι τους αναγκάστηκαν να υποστούν ε, χρονοβόρες ε, δικαστικές διαδικασίες μέχρι να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Νομίζω λοιπόν στην Ευρώπη πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά και αυτά που προσπαθώ να διαβλέψω στην έκθεσή μου είναι η πρόληψη όχι μόνο σε θέματα περιβάλλοντος αλλά και σε θέματα αποκατάστασης και αποζημίωσης ε, ενδεχόμενων ζημιών. Ευχαριστούμε. Επιθυμεί κανείς το λόγο. Κανείς ε, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ε, τροπολογιών είναι η 19η Ιουλίου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνεται λοιπόν. Και τώρα διαπιστώνω ότι έχει έρθει ε, εν πλήρη απαρτία και η νομική υπηρεσία και το Συμβούλιο. Προτείνω λοιπόν ο συνάδελφος κύριος Ράπκα να λάβει το λόγο για το σημείο υπαρθμών 38. Λοιπόν, αναφέρθηκε προηγουμένως η απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Εγώ ε, δεν συμμετείχα σε αυτή τη συζήτηση γιατί... Ε, για να συμμετάσχω σε μια συζήτηση, αυτό σημαίνει ότι έχω δεχθεί την ε, νομιμότητα του Συμβουλίου, κάτι όμως το οποίο δεν δέχομαι. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Τώρα, όσον αφορά ε, τρία θέματα, εκεί πραγματικά έχω ε, ενστάσεις επί της ουσίας. Είναι θέματα που ξεπερνούν τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Καταρχήν, τίτε το θέμα της ουσίας. Νομίζω εχθές η γραμματεία έστειλε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής την πρώτη γνωμοδότηση της νομική μας υπηρεσίας που σημαίνει ότι ε, μπορώ και εγώ να τη χρησιμοποιήσω. Και εσείς την ξέρετε, ούτε και θα ε, κλέψω τίποτα από τη δουλειά του κυρίου Πενέρα. Στο 22 σε στη συνοδευτική επιστολή του κυρίου Πενέρα καθίσταται απόλυτα σαφές ότι η διαγραφή των τριών άρθρων δεν είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο ε, γιατί ε, η διαγραφή, το ενδεχόμενο διαγραφή αντιβαίνει στο 118 που είναι η νομική βάση. Με τη διαγραφή λοιπόν των τριών άρθρων αν υπάρξει αυτή δεν θα υπάρχει και νομική βάση διότι η νομική βάση λέει ότι θέλουμε να έχουμε διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία προστασία και εάν εξαιρεθούν τα άρθρα που παραπέμπουν στην ενιαία προστασία ε, καταπίπτει προφανώς και το άρθρο αυτό. Άρα εδώ δεν μπορούμε να ενδώσουμε. Και αυτό δεν το συζητάμε για πρώτη φορά. Στο Συμβούλιο ε, το ξανασυζητήσαμε αυτό το θέμα στις διαπραγματεύσεις και κατά περίεργο τρόπο, όχι κατά περίεργο, Ούτε και αυτό δεν ισχύει. Εκείνο που ισχύει είναι ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έλαβαν μία απόφαση, αλλά όχι επί της ουσίας, ε, έλαβαν την απόφαση μετά από παζάρι, κατά λέξη παζάρι, όπου υπήρξαν τρεις χώρες που διεκδικούσαν την ενιαία προστασία και για τρεις ολόκληρους το θέμα αυτό αφαιρείτο ή αν θέλετε δεν συμπεριλαμβάνει το καν στη μερίσια διάταξη της Ολομέλειας. Ε, μπορούμε λοιπόν να θεωρούμε ότι είχαμε τύχη που δεν εμφανίστηκαν άλλες πέντε χώρε να διεκδικήσουν την έδρα του ενιαίου δικαστηρίου. Και όλο αυτό το παζάρι οδήγησε σε κάτι όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συγκεκριμένα το άρθρο 15 λέει ότι καμία σχέση ε, δεν έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με νομοθετικές αρμοδιότητες. Και για να το παρακάμψουν αυτό λένε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλή. τι είναι αυτό. Εγώ ξέρω από ανθρώπους του Συμβουλίου που λένε ότι όταν το Συμβούλιο επιλέγει την διατύπωση καλή, κατ' ουσίαν διατάσσει. Και αυτό όμως δεν έχει το δικαίωμα να το πράττει. Κατόπιν τούτου, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, συζητήσαμε και το ε, Συμβούλιο ε, κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων κατέστησε σαφές ότι στηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Στο Συμβούλιο ρωτήσαμε, απευθυνθήκαμε στις νομικές υπηρεσίες και υπάρχει μία απόφαση της νομικής υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την συνάδελφο Βικστρούιμ που κατέθεσε τις σχετικές τροπολογίες. Εγώ λοιπόν ως συγητής παρότι δεν πρόκειται για την δική μου την πολιτική βούληση. παρόλα αυτά είπα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι θα μιλήσουμε για όλα ακόμα και για αυτά ε, που οι συνάλφοι κατέρθεσαν με τη μορφή τροπολογιών. Συζητήσαμε λοιπόν για το θέμα αυτό και κατέστη απόλυτα σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη για λόγους ε, νομικούς και νομιμότητας. Και αυτό λοιπόν το επιβεβαίωσε και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου η θέση ήταν απόλυτα σαφής και αν θυμάστε τις ε, συζητήσεις που κάναμε, δεν υπήρξε καμία διαφωνία από αυτού ε, στις σχέσεις και στις συζητήσεις Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα δηλαδή η απόφαση που λήφθη δεν είναι επί της ουσίας, είναι μια απόφαση μετά από παζάρι και εκείνο που με ενδιαφέρει μένα και πρέπει να το διεκδικήσουμε είναι το εξής. Αν το Συμβούλιο εφαρμόσει αυτά τα οποία αποφάσισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πρέπει να ρωτήσουμε το Συμβούλιο γιατί το κάνει αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει μία επί της αιτιολόγηση πριν γίνει αυτό δεν συζητάμε το Συμβούλιο. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι επιλαμβάνονται του θέματος κάτω από το πρίσμα του ευρωπαϊκού δικαίου, όλοι αυτοί λένε δεν είναι συμβατά αυτά που γίνονται, και ένας ε, λόγος ε, που έχει άμεση σχέση με τον κοινωνού είναι ο εξής. Ο κανονισμός είναι μία ρύθμιση, ρυθμίζει ορισμένα πράγματα. Ε, κατόπιν του πρέπει να λέει τι επιθυμεί να ρυθμίσει. Αν αφαιρέσει κανείς το περιεχόμενο της ρύθμισης, ε, τότε τι νόημα έχει η ρύθμιση. Regulation και μόνο ε, το όνομα στα αγγλικά έχει σχέση με τη ρύθμιση. Ξέρουμε όμως τι κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Πολλοί ήθελαν λοιπόν ε, όχι να κάνουν παζάρι, αλλά να μπουν στην ουσία. Και πάω στο επόμενο θέμα που με ενδιαφέρει. Πίσω από όλα αυτά, δεν λέγονται βέβαια, αλλά κάποια στιγμή πράγματι λέξαν, Θέλουν, διεκδικούν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. θέλουν να αποδυναμώσουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λέω αποδυναμώσουν, ευγενικά το λέω για να μην πω άλλες λέξεις. Όμως αυτό είναι κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο, διότι γνωρίζουμε τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 9-10 όπου μετά από ε, παράκληση του Συμβουλίου συντάχθηκε αυτή η γνωμοδότηση. Το Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να γνωμοδοτήσει για το κατά πόσον το δικαστικό σύστημα της ε, Επιτροπής, που προτείνει η Επιτροπή, είναι συμβατό με, το, ε, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και το δικαστήριο είπε όχι, σε πολλά σημεία δεν είναι συμβατό. Και ένα από αυτά τα σημεία είναι το εξής. Επί της ουσίας, το αποτέλεσμα αυτού υπάρχει πρόταση να αφαιρεθεί το δικαίωμα κατάθεσης προτάσεων. Πολλοί είπαν λοιπόν ότι αυτή είναι μια, ένα τρίκ, μια λύση που τώρα όμως επιλέγεται και τώρα μέσα από τον κανονισμό της ρυθμίσης, δηλαδή προσπαθούν να αφαιρέσουν αρμοδιότητες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω είναι προφανές ε, το τι ακριβώς ε, συμβαίνει. Εδώ όμως πρόκειται για μια ε, πολιτικά αξιοσημείωτη διαδικασία. Και όταν λένε μερικοί ε, ε, θεσμοί, μερικοί συνεργάτες ε, εκτός ε, του θεσμού ότι όλα αυτά όμως δεν θα τα, δεν θα τα σεβαστούμε, αυτά είναι προσωπικές απόψεις. Το να λέει όμως κάτι τέτοιο ένας θεσμός, είτε λέγεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είτε σκέτο Συμβούλιο, αυτό πραγματικά είναι αξιοπερίεργο. Και το καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι να ενισχύει την παραβίαση των συνθήκων, ακριβώς το αντίθετο να την να προστατεύει τις συνθήκες. Πάντως, εάν αφαιρεθούν αρμοδιότητες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, νομίζω θα πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος θεσμός που να προστατεύσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έτσι ώστε να διατηρήσει τις αρμοδιότητες που του έχει εκχωρήσει, το έχουν εκχωρήσει οι συνθήκες. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα και πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό. Και έχω και μία ερώτηση προς τον κύριο Πενέιρα. Πρόκειται για το σημείο υπερθμών 9. Μου είναι απόλυτα σαφές ότι ένα κείμενο αποκτά νομική ισχύ μόνο εφόσον έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους θεσμούς. Σε μας είναι η Ολομέλεια το Συμβούλιο αποφασίζει με τη δική του τη σύνθεση που καθορίζει εκείνο. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τις 2 Δεκεμβρίου υπάρχει μια επιστολή της μόνιμης αντιπροσωπείας εξ ονόματος του Συμβουλίου προς τον πρόεδρο της ε, νομικής επιτροπής όπου αναφέρεται στην επιστολή αυτή ότι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο <coughs> αποφασίσει επί της συμφωνίας τότε δεσμεύεται το Συμβούλιο να εγκρίνει αυτήν την απόφαση λέξη προς λέξη, κυριολεκτικά. Πήραμε λοιπόν αυτήν την επιστολή πριν από λίγο καιρό και κατόπιν τούτου ε, αυτά που αναφέρονται στο σημείο 9 τα κατανοώ ε, από πλευράς νομικής, αλλά εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Και αν δεν υπήρχε και το κάτι άλλο, θα έλεγα να καταργηθούν πλήρως οι τριμερείς αντίσει γιατί πλέον δεν συμβάλλουν σε τίποτα. Και θέλω να προσθέσω και κάτι. Αυτά το ζήσα όλα στο πετσί μου που ήμουν ο βασικός συγητής. Μετά την διασφάλιση της Κορεπέρ εξ του Συμβουλίου και διευκρινίζω, αυτά δεν τα έκανε μόνο η Κορεπέρ. Η Κορεπέρ μίλησε εξ του Συμβουλίου και αναφέρεται στην Επιτροπή κυριολεκτικά for the Council. Έτσι λοιπόν εμείς ε, ψηφίσαμε και ψηφίσαμε κυριολεκτικά όλα αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει. Εγώ, παραδείγματο χάρη, απέσυρα τι ε, τροπολογίε μου ω εισηγητή και σε προτάσεις ε, συναντέλφων που ε, τις θεωρούσα άξιες προ υποστήριξη. Σε τέτοιου είδους προτάσεις είπα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε διότι οι προτάσεις αυτές θα υπονομεύσουν το συμβασμό. Άρα δηλαδή είχαμε μία απόφαση στην Επιτροπή η οποία όμως ελήφθη υπό λάθος πρόσημο ε, κάτω από αρνητικές συνθήκες και πρέπει να πω ότι αν το Συμβούλιο διέγραφε αυτά τα τρία σημεία τότε δεν θα ήταν μόνο θέμα των τριών σημείων αλλά του συνόλου της συμβαστικής πρότασης γιατί δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι συμφωνήσαμε για όλα τα άλλα, για τα τρία αυτά διαφωνούμε, ας τα βγάλουμε απ' έξω, ε, θα εφαρμόσουμε όλα τα άλλα ε, που ε, συμφωνήσαμε. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ σας συστήνω αυτή τη στιγμή να μην διαπραγματευτούμε. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά. Θα πρέπει στη χειρότερη περίπτωση να επανέλθουμε εκεί που ήμασταν σχέδιο έκθεσης και κατάθεση σχεδίου αυτού. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να πω το εξής Είχαμε κάποιες επαφές όπου δεν μιλήσαμε επί της ουσίας, γιατί εγώ αρνούμε να το πράξω αυτό. Μιλήσαμε μόνο επί της διαδικασίας. Και πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους Κύπριους. Ξέρετε γιατί. Γιατί το θέμα αυτό ε, προβλεπόταν στην τελευταία τρίτη της συνεδρίασης της ε, Κορεπέρ και η Κορεπέρα όμως το έβγαλε το θέμα μετά από πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας και γράψανε δίπλα καμία απόφαση. Μιλήσαμε λοιπόν για την περαιτέρω διαδικασία και η Κυπριακή Προεδρία με διαβεβαίωσε Βέβαια μπορεί κανείς να διερωτηθεί τι νόημα έχουν να παίρνει κανείς μια διαβέωση από το Συμβούλιο, έστω και αν αυτή η Κυπριακή Προεδρία. Αλλά εγώ πρέπει να σας πω ότι εντάξει το δέχτηκα, ε, ε, δείχνω εμπιστοσύνη στους ε, Κυπρίους, στην Κυπριακή Προεδρία, που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να ληφθεί απόφαση, ακόμα τουλάχιστον. Και το Συμβούλιο πρέπει να έχει κατά νου ότι αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο ατύχημα που θα μπορούσε να συμβεί ποτέ. Αυτή λοιπόν η κατάσταση. Τις τελευταίες ημέρες ε, είχα έντονη αλληλογραφία και πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση είναι η εξής δεν είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ένα, ένας τρίτος ε, θεσμός. Μερικοί λένε ότι πρέπει κανείς να επιληφθεί του θέματος κάτω από το πρίσμα του ευρωπαϊκού δικαίου. Και όλοι αυτοί λένε, όλα αυτά δεν είναι εφικτά. Εδώ το Συμβούλιο θα αποφασίσει για έναν κανονισμό που είναι άκυρος, χωρίς νομική βάση. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας συστήσω και να παρακαλέσω επί της ουσίας να εξετάσουμε το θέμα περισσότερο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αναβάλλεται η πολιτική μας απόφαση. Όμως Αν υπάρχει μια συγκεκριμένη νομική θέση, τότε διευκολύνεται κατά πολύ η λήψη πολιτικής απόφασης. Γι' αυτό λοιπόν εμένα θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να ε, υπάρξει κάποια τοποθέτηση ε, πάνω σε αυτές εξελίξεις και ίσως μετά το καλοκαίρι ε, μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Και τότε λοιπόν να σκεφτούμε να δούμε τι θα κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Κοιτάξτε κύριε Σιγητά, όσον αφορά την ουσία του κανονισμού, πρέπει να σας πω ότι εδώ επανερχόμεθα σε μια κατάσταση, ε, στην μια κατάσταση που είχαμε και πέρυσι το καλοκαίρι. Δηλαδή, ήταν μια τεράστια διαδικασία. Εμείς ε, κληθήκαμε να διαπραγματευτούμε επ' αυτής. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και μετά, με τη βοήθεια των ε, νομικών υπηρεσιών, ε, συμφωνήσαμε ότι ε, πρέπει να υπάρξει κάποια απόφαση. Τέσσερις έχουν ζητήσει το λόγο. Θέλουμε να ακούσουμε και την Κυπριακή Προεδρία και την νομική υπηρεσία να μιλήσουν καταρχήν οι τέσσερις συνάλφοι και ίσως με τις παρα... παρεμβάσεις να ε, λυθούν τα θέματα. Τα μεταγυρίσει και ο κύριος Πενέρα. Και μετά θα δώσω το λόγο στην Κυπριακή Προεδρία. Να μας πει και εκείνη σύντομα τη δική της θέση. Η κυρία Βίκστρομ χωρίς μικρόφωνο. Κατανοώ απολύτω τον εκνευρισμό των συναδέλφων για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικό το δικό σας κύριε Ράπκάι, που είστε και ο εισηγητής προσπαθείτε να βρείτε ένα συμβιβασμό με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα όσα έκανε το Συμβούλιο μετά από μια συνεδρίαση του εσχής του είδους και κλεισμένων των θυρών ε, που γίνεται ανταλλαγή εμπορευμάτων μεταξύ πρωτευουσών και φυσικά το εθνικό κύρος ακυρώνουν όλες τις θέσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι πονίδιστο αυτό το γεγονός, ήταν πολύ δύσκολο το ζήτημα και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο ε, σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα. Έχουμε μια διεθνή συμφωνία, ένα κανονισμό συναπόφασης και ε, ένα κανονισμό διαβούλευσης και όλα αυτά είναι ενταγμένα σε μια ενισχυμένη συνεργασία προσπαθώντας να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση με τριμερείς συνομιλίες. Αυτό είναι καινοφανές και έχουμε πρόβλημα για τους εξής λόγους. Η πρόταση είναι πολύ επίμαχη, συζητείται εδώ και δεκαετίες και είναι πάρα πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Και όταν καταλήξαμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο για τον νέο κανονισμό για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία, εγώ ήμουν ικανοποιημένη και είχα πιστέψει ότι επιτέλου θα καταλήγαμε σε συμφωνία. Δεν με ικανοποιούσαν βέβαια όλε οι πτυχέ τη, όπω θα θυμούνται και οι συνάδελφοι. Είχα προτείνει κάποια στοιχεία τα οποία ε, δεν ελήφθησαν υπόψη στη συμφωνία με το Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά εγώ και οι φιλελεύθεροι ε, στο Κοινοβούλιο εξακολούθησαν να υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Όμως ε, αυτή η μεταμεσανίκτια συμφωνία ε, ουσιαστικά ε, υλοποίησε και έφτασε σε κάτι το οποίο εγώ επί της ουσίας εγκρίνω, αλλά ήταν η διαγραφή του άρθρου 6 και 8 και καταλαβαίνω ότι πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να έχουμε καταλήξει και στο αντίθετο αποτέλεσμα. Κανεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμού συμπεριλαμβανομένε, δεν θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένοι από την πρόταση αυτή, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουμε για την ουσία του ζητήματο. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει ε, να είναι πολύ ε, προσεκτικό και δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να προδικάσει την συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι ε, πώς θα καταλήξουμε σε συμφωνία επί της ουσίας εμείς θα είχαμε υποστηρίξει αυτό το ευρωπαϊκό δίπλωμα ε, ευρεσιτεχνίας και με τα άρθρα 6, 7 και 8 παρά το γεγονός ότι δεν ήταν η αρχική μας πρόθεση. Αυτό το είχαμε ε, δείξει και με την ψηφοφορία μας εδώ στην Επιτροπή το Δεκέμβριο. Επί της ουσίας όμως θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε και ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χωρίς αυτά τα άρθρα διότι εγώ ζητούσα να διαγραφούν από τον κανονισμό σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εδώ στην Επιτροπή μας όταν το συζητούσαμε. Δεν θεωρώ ότι σήμερα θα πρέπει να επανέλθω στην ουσία για το κατά πόσον είμαι υπέρ ή κατά τη διαγραφή των, της διαγραφής των άρθρων, θα πρέπει να γίνει μια πολύ πιο διεξοδική συζήτηση επί του ζητήματος. Θα μπορούσα κάλλιστα βέβαια να το συζητήσω αργότερα, αλλά αυτό που έχει περισσότερη σημασία κατ' εμέ είναι να προσπαθήσουμε να εργαστούμε με ευέλικτο τρόπο και να είμαστε και δημιουργικοί για να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση και σύντομα μάλιστα η κοινή συμφωνία με το Συμφωλείο είναι ο τελικός μας στόχος. Και αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει εκνευρισμός, αλλά κάνω έκκληση προς όλους στην Επιτροπή μας δεν θα πρέπει ε, να δείξουμε την απογοήτευσή μας, διότι μας ενδιαφέρουν οι πολίτες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη και όλοι όσοι ε, θέλουν να καταθέσουν διπλώματα ευρεσιτεχνίες. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για αποτυχία αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη διανύει κρίση και εμείς έχουμε εκλεγεί για να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα της Ευρώπης. Δεν θα είναι βέβαια εύκολο, αλλά ελπίζω ότι από κοινού θα μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο για να λήξει επιτέλους αυτό το το θέμα. Διότι αυτό πρέπει να γίνει. Όπω είπε και ο συνάδελφο Ραπκάη, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τι καλοκαιρινέ διακοπέ ε, ο ενίδη περισυλλογή και να επανέλθουμε το Σεπτέμβριο με περισσότερη ενέργεια και ίσω να είμαστε και λίγο πιο εφάνταστοι και να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα δια μια. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριο Πασκουάλ Ντεγκράντε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι γνωστό τη σπάση ποια θέση έχει η Ισπανική Αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και είναι γνωστό ότι και οι σοσιαλιστές συντάσσονται με τη θέση των Ισπανών στο ΕΛΚ. Και οι Ισπανοί σοσιαλιστές, συγγνώμη. Είμαστε κατά τη συμφωνία αυτή και δεν είμαστε κατά επειδή ε, δημιουργείται ένα ενιαίο ε, δίπλωμα ευαισθητεχνίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Αλλά υπήρξαν ε, πολλές ε, ελλείψεις και μάλιστα ασκήσαμε και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπήρχαν και προσφυγές στο δικαστήριο. Και μάλιστα φαίνεται ότι παραγωνίστηκαν εσκεμένα σημαντικές γλώσσες όπως ε, η Ισπανική που τη μιλούν 50 ε, εκατομμύρια Ισπανόφωνοι. Συγγνώμη, ε, πολύ περισσότεροι Ισπανόφωνοι στον κόσμο. Θα ήταν πολύ κοινικό να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε βέβαια μειοψηφία στη θέση αυτή και το γεγονό ότι το Συμβούλιο ομόφωνα έλαβε θέση και κατήργησε τα άρθρα 6-8 του ουσιαστικού κανονισμού για το ενιαίο δίπλωμα βεστεχνία μα δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Όπω μα είπε η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτή η κατάργηση στερεί περιεχομένου το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα και άρα δεν ε, έχει νόημα η νομική βάση που επιλέγεται για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η νομική βάση ούτως ή άλλως φαίνεται αυτή αντιβαίνει στην υλοποίηση της ισοενιαίας αγοράς. Μα ανησυχεί το γεγονό ότι η συζήτηση για την κεντρική έδρα του δικαστηρίου κράτησε έξι μήνες, πολύ περισσότερο από την ίδια τη συζήτηση για το περιεχόμενο του ενιαίου διπλώματο ευαισθητεχνία. Είναι πραγματικά λυπηρό και μάλιστα αυτοί, οι διαξυφισμοί για την έδρα δεν εξυπηρετούν κανένα παρά μόνο κάποια εθνικά συμφέροντα και σίγουρα δεν μα περιποιούν τιμή. Το αντίθετο. Φύγουν το κύρος και την έγκλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε την ε, νομική υπηρεσία στις 18 και ε, ε, θα ακούσουμε και τη συζήτηση 18 και 19 Ιουλίου. Θα δούμε ποια θα είναι η γνώμη, η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και η προτάση για να ξεφύγουμε από αυτό το χάος και το αδιέξοδο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον Γενικό Διευθυντή της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να του δώσω το λόγο αργότερα να μας παρουσιάσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Μασίπ, θα ήθελα να συμφωνήσω 100% με την πολύ εύγλωτη και εύστοχη ομιλία του κυρίου Δεγράντες Πασκάλ, του εκπροσώπου του ΕΛΚ, της Ισπανικής Αντιπροσωπείας του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Μπαλτασάρε. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε το θέμα καταρχάς βάσει των προτεραιοτήτων μας. Καταρχάς η πρώτη παρατήρηση είναι ότι αυτό το οποίο συνέβη είναι ένα πολύ κακό πολιτικό προηγούμενο. Δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα και κανένα δικαίωμα να ανακατεύεται ε, το δικαστήριο σε μια νομοθετική διαδικασία την οποία προχωρά, ε, ε, προχωρούν οι δύο συνομοθέτες. Δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών Στη διάρκεια της πολωνικής προεδρίας είχαμε καταλήξει σε μια συνεννόηση. Πρέπει να πω ότι το Κοινοβούλιο είχε δείξει μεγάλη αίσθηση ρεαλισμού και είχε δεχτεί μια σειρά από προϋποθέσεις που είχαν προέρθει από κάποια κράτη-μέλη και πραγματικά ειλικρινώς η παρέμβαση η οποία έγινε τις προηγούμενες ημέρες δεν έχει καταρχάς καμία νομική υπόσταση. Πέραν αυτού, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε μια λύση και ότι οι βασικές προϋποθέσεις είναι καταρχάς ο σεβασμός του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά δεύτερον μια διάφανη διαδικασία, σαφής, η οποία θα γίνει με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Εν κατακλείδη, εμείς πάντα ήμασταν ρεαλιστές και θέλαμε να καταλήξουμε σε συμπέρασμα, διότι εδώ και 30 χρόνια περιμένουμε ένα αποτέλεσμα και ο όλος ο βιομηχανικός κόσμος και ο κόσμος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να μας ζητάει να καταλήξουμε πλέον σε αυτό το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ε, το οποίο παρακολύουν οι εγωισμοί των κρατών μελών και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας καθοδόν. Ε, χάθηκαν πάρα πολλές τροπολογίες ε, στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Είχαμε καταλήξει σε κάποιο σημείο στο οποίο θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και έχουμε το καθήκον να συνεννοηθούμε και μετά από αυτή την παρέμβαση η οποία τροποποιεί ουσιαστικά ε, τρία πολύ σημαντικά άρθρα. Η σημασία του έργου αυτού είναι πάρα πολύ μεγάλη και πραγματικά ειλικρινά πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος εδώ να γίνονται ε, γλωσσικές ε, μάθες. Καταλαβαίνω τη θέση της ισπανικής αντιπροσωπείας, καταλαβαίνω και τη θέση της ιταλικής κυβέρνησης, αλλά εγώ είμαι αντίθετος, διότι το 90% των ιταλικών επιχειρήσεων καταθέτουν αιτήματα ε, για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα αγγλικά, το 2% στα γαλλικά και το 1% στα γερμανικά. Σημαίνει ότι το γλωσσικό ζήτημα δεν είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί κόσμος των επιχειρήσεων ούτως ή άλλως έχει ενία γλώσσα στην Ευρώπη. Αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρηθεί αυτή η αλλως εχει μια γλωσσα στην ευρωπη αυτο που εχει παγκοσμίω και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να γίνονται εδώ πέρα αυτές οι διαμάχες ε, για το σε ποια γλώσσα θα γίνει τι. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει αυτό το έργο ε, διότι είναι θεμελιώδης σημασία και για το σύστημα καινοτομία, το οποίο ζητούν ε, αρκετέ πλευρές και για να καταφέρουμε με ακρίβεια να καταλήξουμε επιτέλους σε ένα συμπέρασμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λίχτεμπεργκερ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω πλήρως με την ανάλυση που μας έκανε ο συνάδελφος Σαράπ Όντως διαπιστώνουμε ότι ένας ολόκληρος κανονισμός εκενώθηκε περιεχομένου, απογυμνώθηκε από το συστικά του σημεία, κάτι που αντιβαίνει στις αρχικές μας προσδοκίες και στόχους. Δηλαδή, την αναζήτηση του κοινού παρανομαστή για το θέμα αυτό στην Ευρώπη. Δεν κατέστη δυνατό, δεν πρόκειται να επαναλάβω τα επιχειρήματα που ακούσαμε. Το Συμβούλιο μας κατέκλυσε με πληροφορίες και μας προσπάθησε να μας πείσει για τη σπουδαιότητα αυτού του θέματος. Ναι, μιλήσαμε για τα παζαρέματα. Όντως έγιναν παζαρέματα που δυστυχώς απογύμνωσαν την πρόταση από το περιεχόμενό της. Γι' αυτό και δεν έχει νόημα πια να συνεχίσουμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε να κινήσουμε και πάλι τη διαδικασία, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε εκ του μηδενός και πάλι, γιατί επαναλαμβάνω, εκενώθηκε περιεχομένου η πρόταση αυτή με την κατάργηση των άρθρων. Οπότε και η άλλη πρόταση, η εναλλακτική, δημιουργεί τεράστιες αβεβαιότητες και αντιβαίνει στην ασφάλεια του δικαίου. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, πολλές απορίες, ενώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταλήξουμε σε ένα ουσιαστικό, γνήσιο, ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία στην Ευρώπη. Και το γλωσσικό ζήτημα δεν είναι πια το πιο αποφασιστικό και το πιο κρίσιμο. Το αποφασιστικό σημείο στο θέμα αυτό είναι αν κάποιο που θέλει να κατοχυρώσει ένα δίπλωμα ευρυστεχνία θα έχει μια νομική ασφάλεια με την κατοχύρωση αυτή στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Θα εξασφαλίσουμε αυτή τη νομική ασφάλεια που θα ανταποκρίνεται στους στόχους του κατόχου του διπλώματος ευρυστεχνίας. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσω και τη γνώμη της Κυπριακής Προεδρίας, τη γνώμη του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Τι θα πούμε στους ανθρώπους που θέλουν ε, και βάλουν έτοιμα για ένα νέο δίπλωμα ευρυστεχνίας. Θα τους εξασφαλίσουμε μια γνήσια και πλήρη νομική ασφάλεια ή μόνο μια μερική ασφάλεια δικαίου. Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για το σημείο αυτό και αν δεν εκφράσουμε ενιαία φωνή, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε και πάλι εκ του μηδενό όπω πρότεινε ο κύριο Ραπκάη. Που σημαίνει ότι και πάλι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε για τα ποιο είναι τα κέρια σημεία τη πρόταση και για ποια σημεία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Επίσης θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιος ενδιαφέρεται για τα σημεία αυτά, ποιος θέλει να τα προωθήσει και ποιος έχει συμφέρον να αποτελματωθεί η συζήτηση και να μπλοκαριστεί. Δεν θέλω να με θεωρούν ανόητη. Δεν συμφώνησα, ούτε πρόκειται να συμφωνήσω για σημεία που στη συνέχεια παραγωνίζονται ή χρησιμοποιούνται με στρεβλό τρόπο. Δεν θέλω να είμαι... Ε, ε, να μην συνεργαστώ, δεν θέλω να μη δείξω επικοδομητική συνεργασία, αλλά ούτε θέλω να με περνάει και για χαζή. Έχουμε πολύ ε, σημαντικά θέματα. Έχουμε εδώ την τριπλή έδρα. Για την έδρα είπαμε θα πρέπει να περιορίσουμε ε, την τριπλή έδρα και τώρα βλέπουμε ότι τρία κράτη-μέλη διαγωνίζονται για την έδρα. Γιατί να μιλούμε για τον αριθμό των εδρών και να περιοριζόμαστε σε τρει, α πούμε από την αρχή ότι το δικαστήριο θα έχει 27 έδρε, άμα θέλετε, για να ικανοποιηθούν όλοι. Βλέπω εδώ και μία πολιτική απειλή υπάρχει κίνδυνος να ε, αφήσουμε και τη σύμβαση του ανθρωπίνου δικαιωμάτων γιατί θα μπει η διαδικασία στη δική της δυναμική και κάθε έδρα θα είναι δικαιωμένη με τον τρόπο που επιθυμεί. Τι θα γίνει με όλες αυτές τις αντιφάσεις που δημιουργήθηκαν, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ναι, ωραία να λέμε ότι θα πρέπει να βρούμε νέες διεξόδους για τους ειδικευμένους δικηγόρους σε θέματα διπλωμάτων ευρυστεχνίας, αλλά θα πρέπει κάτι τέτοιο να γίνεται εις βάρος του εμπορίου δεν φταίει η διαδικασία γι' αυτό, αλλά η στάση του συμβολίου, η συμβολίου ήταν ανεύθυνη κυρίως. Um, Θα ήθελα να συμφωνήσω με τα όσα είπε η συνάδελφος κυρία Wickstrom είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε σε ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνία στο συντομότερο δυνατόν, διότι θα είναι προ όφελο ε, των επιχειρήσεων και των μεγάλων και των μικρομεσαίων και φυσικά θα βοηθήσει και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ενώπιον των ΗΠΑ και ενώπιον ε, τη Ασία φυσικά. Ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διάρκεια του θέρου με του νομικού εμπειρογνώμονε στον τομέα, ώστε να ε, είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι νομικά ασφαλέ το δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Ο κύριος Καρίμ. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω και τη δική μας τη θέση. Καταρχάς, για τα άρθρα 6 έως 8. Εγώ προσωπικώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαγραφούν τα άρθρα αυτά από τις διατάξεις. Δεν θεωρώ ότι η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δημιουργεί διαφορετικό ε, προηγούμενο βάσει και των καθυστερήσεων που είχαμε ε, με το φόρτο εργασίας που έχουν αυτή τη στιγμή ήταν πρόοδος. Ούτως ή άλλως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, ένα εξειδικευμένο σύστημα το οποίο θα ασχολείται με συγκεκριμένα ζητήματα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα, για να δούμε κάποια από τα βασικά ζητήματα. Συμφωνώ με την απογοήτευση των συναδέλφων ε, για τον αριθμό των εδρών ε, που θα είναι διαθέσιμες και όλο το γλωσσικό ζήτημα. Αλλά Κύριε Πρόεδρε, στο κάτω-κάτω της γραφής Ευρώπη είμαστε και κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα. Έχουμε πάρει κάτι απόλυτα λογικά και έχουμε καταφέρει να το ε, διαλύσουμε ένα προς ένα και να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα κοιτούν οι πολίτες μας και θα λένε τι στο καλό κάνατε. Πραγματικά θα μπορούσαμε να τους είχαμε πει ότι θα έχουμε μια έδρα στη Φραγκφούρτη που θα μιλούν αγγλικά, μια στο Παρίσι που θα μιλούν γερμανικά και έχουμε και μια στο Λονδίνο όπου θα μιλούν γαλλικά. Και ε, θα υπάρχει και μια υφέρπουσα γλώσσα και ο καθένας θα μπορεί να έρθει και να μιλήσει ισπανικά όποτε τον βολεύει. Ε. Νομίζω ότι ε, τελικά τα ε, υπερτιμάτε λιγάκι. Έτσι κι αλλιώ ε, τα περισσότερα ρυθμίζονται σε περιφερειακό επίπεδο. Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου που θα είναι τελικά η έντρα. Νομίζω ότι τα τοπικά δικαστήρια είναι εκείνα τα οποία τελικά αποφασίζουν. Εκεί έχουμε του δικηγόρου που ασχολούνται με θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Α μην κοροϊδευόμαστε. Οι άνθρωποι αυτοί θα προσπαθήσουν να εγκατασταθούν εκεί κοντά που θα είναι και το δικαστήριο. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Πενέρα. Εχθές στις συζητήσεις που είχα με τους ε, Βρετανούς εμπειρογνώμονες μου είπαν ότι το άρθρο 3 αρκεί και περισσεύει για να ε, αιτιολογεί τη νομική βάση του 118. Μήπως μπορείτε να τοποθετηθείτε λιγάκι από αυτού, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δεν πρόκειται να αναφερθώ στο ουσιαστικό περιεχόμενο της γνωμάτευση νομικής υπηρεσίας, γιατί σας μοιράσαμε το κείμενο της γνωμοδότησής μας, είναι σαφέστατη. Εμείς πιστεύουμε ότι η διαγραφή των άρθρων 6-8 ε, αφορά ουσιαστικά σημεία της πρότασης και διερωτώ με... Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θέλει ένα στόχο και ένα περιεχόμενο για κάθε νομική πράξη. Υπάρχει βέβαια περιεχόμενο σε αυτή την ε, πράξη, αλλά δεν υπάρχει πια στόχος έχουμε μία νομοθετική πράξη που στερείται αντικειμένο. Δεν υπάρχει πια αντικείμενο σε αυτή την πράξη. Αφαιρέθηκε το αντικείμενο, το ίδιο το αντικείμενο, το, ο ίδιος ο στόχος από την νομοθετική αυτή πράξη. Τώρα, αν το άρθρο 3 αρκεί από μόνο του, μπορεί κανείς να γίνει λιτός και απέριτος και μινιμαλιστής. Ε, σίγουρα το απόγειο της, ε, του μινιμαλισμού είναι η σιωπή το, απόγειο της α, ε, σύνθετης ε, ομιλίας είναι η σιωπή. Είχαμε 25-26 σελίδες ε, γνωμάτευση. Να εμείνουμε στο άρθρο 3. Πάντα κάποιος θα βεβαιωθεί που θα πει ότι αρκεί το άρθρο 3, άλλος θα πει αρκεί το άρθρο 9. Πάντως το θέμα είναι ότι αν διαγραφούν αυτά τα τρία σημαντικά άρθρα, 6, 7 και 8, ουσιαστικά ακυρώνεται η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου και πλήττουμε την ίδια την αξία του διπλώματος ευρυστεχνίας ως ομοιόμορφου και ενιαίου διπλώματος. Τώρα σε ό,τι αφορά την ακολουθητέα πρακτική, το αναφέρουμε στο σημείο 9 της γνωμοδότησης με το θέμα αυτό. Οι προπαρασκευαστικές φάσεις, τριμερής διάλογος και η μεθοδολογία που θέτησε στη συνεργασία του Συμβούλιο και Κοινοβούλιο για να καταλήξουν σε απόφαση σε πρώτη ανάγνωση είναι διαδικασίες που δεν αποκλίνουν από τη συνθήκη. Και μάλιστα είναι πολύ νοχλητικό που η σιωπηρή συμφωνία ή έστω και τη δηλωμένη συμφωνία του Συμβουλίου που ε, οδήγησε την ε, νομική υπηρεσία στην αγνομοδότηση της ε, Καλόπιστα, ελπίζοντα ότι αυτή ήταν η βούληση του Συμβουλίου να ολοκληρωθεί το θέμα σε πρώτη ανάγνωση. Και το θέμα είναι τι θα κάνετε εσεί με τη δική σα έκθεση. Γιατί τεχνικά υπάρχει η δική σας έκθεση. Θα πρέπει να βρεθεί ένα άρθρο του κανονισμού που να επιτρέπει ε, να επανέλθετε στην έκθεση χωρίς να την καταθέσετε στην Ολομέλη Γιατί πλέον στερείται αντικειμένου και στόχου αυτή η πρόταση. Τώρα, Ποιο είναι το αρνητικό. Το, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει νομοθετική αρμοδιότητα. Προτείνει αλλά δεν μπορεί να παρέμβει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τυπικό ελάττωμα στην περίπτωση αυτή, διαδικαστικό ελάττωμα. Όλη η διαδικασία που εφαρμόστηκε εδώ και χρόνια για τις πρώτες αναγνώσεις, για τις συμφωνίες, τις γραπτές ε, από το Συμβούλιο ε, και την τήρηση των συμφωνηθέντων θα πρέπει να ακολουθηθεί. Το Κοινοβούλιο έχει συμφέρον να ακολουθήσει αυτή την πρακτική. Αλλά εδώ έγινε μια παράκαμψη. Ε, βραχικυκλώθηκε το κείμενο, βραχικυκλώθηκε η διαδικασία. Έχουν μείνει στάχτες μόνο από το κείμενο. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια δεσμευτική αξία. Υπάρχει μια δεσμευτική αξία στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας αλλά η πάγια νομολογία του δικαστηρίου δεν αμφισβητεί τη δική σας απόφαση. Πάντως ε, ε, είναι έμεση η υποχρέωση του Συμβουλίου θα πρέπει να περάσει στη δεύτερη ανάγνωση. Και ακόμη και αν το Κοινοβούλιο έδωσε τη θέση του, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ανα πάσα στιγμή να ανακαλέσει ε, το κείμενο της, την νομοθετική της πρόταση. Αυτό το ξεχνούμε. Αν, θεωρούμε ότι, αν θεωρεί ότι αελιώθηκε η νομοθετική πράξη, μπορεί καλή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της, ανά πάσα στιγμή, σε επίπεδο συνομιλιών στο Συμβούλιο στην πρώτη ανάγνωση. Αυτά. Αν θέλετε ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις να απαντήσω. Δεν έχει νόημα τώρα να συνεχίσω. Νομίζω ότι είναι ε, προφανής η θέση μας αυτή τη γνωμοδότηση που σας δώσαμε. Θα συνεχίσουμε πάντως ε, τη συνεργασία και με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου, προσπαθώντας να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα διεξόδου σε αυτή τη μέχρι στιγμή ατυχή εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Γενική, η Κομισιόν, Γενική Διεύθυνση, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικός ε, δεδομένης και της συζήτησης ε, που μόλις ακούσαμε. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία αυτού του ζητήματος ε, που μας έχουν κάνει να μετανιώσουμε στη διάρκεια των ετών και ίσως το πιο σημαντικό εξ αυτών είναι η καθυστέρηση στην τελική συμφωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να υπενθυμίσω ε, πόσο σημαντικό είναι να καταλήξουμε σε τελική συμφωνία για την ενιαία αγορά, για τις επιχειρήσεις, για τους επενδυτές και φυσικά για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρειαστούμε, χρειαστήκαμε ανέκαθεν τη συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων για να καταλήξουμε στο στόχο να έχουμε το πρώτο ενιαίο ε, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τον Απρίλιο του 2014. Σημειώνουμε φυσικά τα όσα συνέβησαν στο ε, Συμβούλιο της Προάλλες, ε, τα ξημερώματα ή το βράδυ και λαμβάνουμε υπόψη και το έγγραφο από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου, το οποίο μόλις λάβαμε και λέει ότι η διαγραφή των άρθρων 6 έως 8 διακυβεύουν ε, τα όσα λέει το άρθρο 118 και διακυβεύεται η νομική βάση του κειμένου. Ε, είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να ε, επιλύσουν όλα τα εκκρεμή νομικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ακούσουμε την Κυπριακή Προεδρία. Δεν ξέρω ποιος από εσά θέλει το λόγο εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας. Thank Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας πω ότι παρακολούθησα τη συζήτηση ιδιαίτερα προσεκτικά όσα ακούστηκαν λαμβάνονται δεόντως υπόψη και φυσικά θα τα μεταφέρουμε στο Συμβούλιο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ως Προεδρία συνειδητοποιούμε πλώρε ε, πόσο ε, σημαντικό είναι να υπάρχει ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνία, ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια. Εξακολουθούμε στη δέσμευσή μας να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Έχει γίνει πολλή δουλειά για το ζήτημα αυτό εδώ και αρκετά χρόνια και δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Φοβούμεθα ότι ε, εάν δεν τα καταφέρουμε και χαθεί η ευκαιρία αυτή, θα χρειαστούν ίσως πολλά χρόνια πριν καταλήξουμε ε, σε συμφωνία για το θέμα αυτό. Πώς έχει τώρα το θέμα στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα για το Συμβούλιο τουλάχιστον ήταν ότι χρειαζόμασταν ένα συμβιβασμό για το θέμα της έδρας. Και ο συμβιβασμός επετεύχθη στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με μία πρόταση τη διαγραφή των άρθρων 6 έως 8 από τον κανονισμό. Κατανοούμε τον εκνευρισμό ε, και τη δυσαρέσκεια που έχει δημιουργήσει αυτή η απόφαση. Είχαμε θεωρήσει ότι αυτό που είχε σημασία είναι να έχουμε όλοι τον κατάλληλο χρόνο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να σκεφτούμε ξανά το ζήτημα και να το συζητήσουμε εκ νέου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Εν τω μεταξύ, αν κατάλαβα καλά, θα ε, υπάρξει και άλλη νομική γνωμοδότηση για συζήτηση από πλευρά σας το Σεπτέμβριο το Συμβούλιο ε, ακολουθεί αντίστοιχη άγουσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το, ε, το ίδιο και ελπίζω στις αρχές Σεπτεμβρίου να είμαστε σε θέση να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι με τις γνωμοδοτήσεις των νομικών υπηρεσιών ενώπιών μας και επί τη βάση αυτών των γνωμοδοτήσεων να μπορέσουμε να λάβουμε τις απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις οι οποίες ε, θα μας οδηγήσουν ε, στο ε, επιτυχές αποτέλεσμα αφού προχωρήσει το ζήτημα. Αυτά είχα να σας πω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρέσβη, άλλοι δύο έχουν ζητήσει το λόγο και στο τέλος θα δώσω το λόγο στον κύριο Ράπκαη. Ρίξτρομ, Λίχτενμπεργκ και Ράπκαη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν είχα την πρόθεση να αναφερθώ σε αυτά τα τρία άρθρα. Αλλά μια και όλοι οι υπόλοιποι μίλησαν για αυτά, θα σα δώσω και εγώ τη γνώμη μου για την πρόταση διαγραφή των τριών άρθρων. Το πρόβλημα τη συμπερίληψη των άρθρων 6, 7 και 8 στον κανονισμό είναι ότι μετατρέπονται έτσι σε ευρωπαϊκό δίκαιο, κάτι που δίνει ε, δυνατότητα και προδικαστικών και παραπομπών προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ερμηνεία αυτών των άρθρων κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον κόστο πιο χρονοβόρε διαδικασίες για όλους τους ενδιαφερόμενους, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Άλλωστε, ε, έχουμε νέο ειδικό δικαστήριο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Γιατί να κάνουμε ειδήμονα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που θα καλείται να, με προδικαστικά ερωτήματα να ερμηνεύσει τα άρθρα αυτά. Χρειαζόμαστε πιο ουσιαστικό δίκαιο ε, στη, στο ουσιαστικό δίκαιο, περισσότερες διατάξεις ε, για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Και είχα πολλά mail από δικηγόρους, από οργανώσεις επιχειρήσεων, από πανεπιστημιακούς ε, και από δικαστές για διπλώ, ειδικούς στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Όλοι ομόφωνα τάχθηκαν υπέρ της διαγραφής αυτών των τριών άρθρων. Είναι κατά των τριών άρθρων. Όλοι αυτοί. Γι' αυτό και εγώ είμαι υπέρ της διαγραφής των τριών άρθρων. Και το είπα αυτό στη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου, αλλά δυστυχώς δεν ακούστηκε φωνή μου. Απέτυχα. Τώρα που θα ε, χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρόνο για να ξανασκεφτούμε τα θέματα και να προβληματιστούμε, θα πρέπει να, να προβληματιστούμε. Ποιοι είμαστε εμείς για να ε, λάβουμε διαφορετική θέση από τόσους ειδικού, δικαστές, πανεπιστημιακούς, νομικούς που τάσσονται υπέρ της διαγραφής των τριών άρθρων. Ναι μεν είμαστε εδώ για να εκπροσωπούμε τους πολίτες, αλλά είμαστε εδώ για να ακούμε και όλα τους πολίτες και τους ειδικού και να μαθαίνουμε. Θα ξανάρθουμε το Σεπτέμβριο για να ακούσουμε, να μάθουμε, να προσαρμοστούμε και να συνεχίσουμε την πορεία μας για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ε, τον υπάρχουν τόσα πολλά ε, email, αυτό μάλλον είναι ένας κακός ιονός. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω μπερδευτεί με όλα αυτά που έχουν λεχθεί εδώ, κυρίως με τις τελευταίες παρατηρήσεις. Διότι ο δικός μας ο ρόλος δεν είναι μόνο να ακούμε και να μαθαίνουμε, αλλά και να αποφασίζουμε. Και σε τελική ανάλυση ε, να τηρούμε, να παραμένουμε πιστοί στις αποφάσεις μας. Έστω και αν ε, είμαστε πρόθυμοι για συμβασμού. Απευθύνομαι στην Κομισιόν. Πολύ καλή και διπλωματική η τοποθέτησή σα. Αλλά ξέρετε κάτι, με τη διπλωματία και μόνο δεν μπορεί κανεί να προχωρήσει. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση που στο Συμβούλιο διατηρηθούν αυτά τα τρία άρθρα. Ερωτώ λοιπόν, η Κομισιόν είναι πρόθυμη να αποσύρει την πρότασή της για να ε, ξεκινήσει από την αρχή ή όχι. Γιατί δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να συνεχίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Ε, κοιτάξτε, υπάρχουν διάμεσα και δύο αναγνώσεις και μία διαπραγμάτευση. Μην το ξεχνάτε. Συνάλφος Έγκστορμ. Η κυρία Βίκστρομ ε, είπε κάτι που με εξέπληξε. Στόχος μας δεν είναι ε, να γίνει αυτή η νομοθεσία για να ικανοποιήσουμε τους ε, δικαστές που θα ασχολούνται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα δίπλωμα το οποίο θα είναι όσο καλύτερο για τις επιχειρήσεις και την καινοτομία και ήλπιζα να συμφωνούμε όλοι από αυτού. Δεν γίνεται προ όφελο των δικηγόρων, των νομικών και των δικαστών που θα ασχολούνται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Είναι προ όφελο τη καινοτομία στην Ευρώπη. Εμεί ω πράσινοι υποστηρίζουμε πάντοτε ότι θα πρέπει να υπάρχει νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνία, το οποίο θα εισαχθεί καταλήλω και στι ε, ε, δικαστικές και στις νομικές δομές στην Ευρώπη διότι ερίζουν οι απόψεις για το ποιο θα είναι το τέλειο ε, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και το σύστημά του αλλά πρέπει να συμφωνούμε όλοι στο γεγονός ότι είναι πολιτική απόφαση. Είναι ένα από τα λίγα πολιτικά μέσα που έχουμε εμείς ως πολιτικοί για να επηρεάσουμε την καινοτομία. Ε, ναι, θα ήταν ευπρόσδεκτο ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία αν ήταν ένα ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία όπω πρέπει με τον κατάλληλο δικαστικό και νομικό έλεγχο. Στόχο όμω του συστήματο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία είναι να είναι ένα σύστημα το οποίο θα είναι καλό για την καινοτομία, όχι να είναι καλό για του νομικού που θα ασχολούνται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Ευχαριστώ. Η κυρία Λίχτενμπεργκερ υπέβαλε μια συγκεκριμένη ερώτηση προς την Επιτροπή. Ίσως μπορεί να απαντήσει η Επιτροπή και μετά ο συνάδελφος κ. Ραπκάη. Ευχαριστώ. Στόχος μας εξακολουθεί να είναι να βοηθήσουμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε συμφωνία. Προς το παρόν δεν θέλω να ξεκινήσω οικοτολογίες και υποθέσεις για το τι θα κάνει η Επιτροπή με την πρόταση της. Η πρόταση είναι επιτάπητος, έχει ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία συνεχίζεται και ευελπιστούμε ότι Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Και όπως είπαμε και προηγουμένω, η Επιτροπή θα, βοηθήσει, θα προσπαθήσει να βοηθήσει να διευκολύνει την κατάληξη συμφωνίας. Πολύ διπλωματική απάντηση. Ναι. Κοιτάξτε, θα ήθελα η Κομισιό να δείξει ε, λίγο μεγαλύτερη στράτευση για τη δική της την πρόταση, να την υπερασπιστεί. Τι ήταν αυτό, τίποτα δεν είπε. Μα δεν σκέφτηκε ο Μισιόν ότι πρέπει εδώ να υπεραμεινθεί τη δική τη της πρότασης. Δεύτερον, αυτό που είπε τώρα στο τέλος ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος τελικά κατέληξε στο ότι θα πρέπει να καταλήξουμε το στομό των δυνατών σε μια συμφωνία. Μα αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, έχουμε μια συμφωνία που είναι 9 μηνών. Όποιος λοιπόν μας λέει ότι θα πρέπει το των δυνατόν να καταλήξουμε συμφωνία, ε, φαίνεται ότι την τελευταία χρονιά κοιμόταν βαθιά τον ύπνο του δικαίου ή αν δεν το έκανε αυτό, θέλει να μας εξαπατήσει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχει συμφωνία και πλέον εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στο Συμβούλιο να επανέλθει σε εκείνο στο οποίο έχουμε συμφωνήσει. Όχι στο πειρά, αλλά με μια επιστολή. Περί αυτού πρόκειται. Και εγώ παρουσίασα την άποψή μου και θέλω παρόλα αυτά να πω δύο θέματα. Το πρώτο που θέλω να πω ε, βασικά έχει σχέση με αυτά που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή το Συμβούλιο για 10 ολόκληρα χρόνια εμπόδισε το να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνές και τώρα κάνει το ίδιο. Το λέω ξεκάθαρα. Αν δεν έχουμε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας γι' αυτό θα φταίει μόνο το Συμβούλιο, κανείς άλλο, ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε κανείς άλλο το ε, Συμβούλιο καθυστερεί συνεχώς. Ε, το λέω αυτό για να ε, προλάβω τις φήμες, γιατί μερικοί θα λένε ότι μα ενδώστε και εσείς λίγο. Όχι, όχι, όχι, αυτά δεν γίνονται. Ευθύνη φέρει το Συμβούλιο, ξεκάθαρα και οποιαδήποτε γνωμοδότηση ε, θα ε, κάνω από τώρα και στο μέλλον θα το αναφέρω συνέχεια. Το Συμβούλιο φταίει που δεν υπάρχει ευρωπαϊκό δίπλωμα Ευρωστηχνής. Και μια φιλική τώρα παρατήρηση προς τη Σεσίλια. Πριν από μερικούς μήνες το έχει ξαναπεί. Ε, να σου το πω τώρα και εγώ ξεκάθαρα. Όταν ε, ρωτάς, μα ποιοι είμαστε, <laughs> να σου πω ποιοι είμαστε. Είμαστε κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε το κοινοβούλιο. Και εμείς είμαστε οι μόνοι οι οποίοι Λόγω της εκλογής μας ε, είμαστε νομιμοποιημένοι να θεσπίζουμε νόμους. Ε, νόμους δεν θεσπίζουν οι ε, δικηγόροι των διπλωμάτων. Το δικό μας το καθήκον δεν είναι να διασφαλίζουμε τη δουλειά των δικηγόρων. Και ξέρεις, και εγώ πήρα πολλές email που θέλουν να διαγράψουν το 6 μέχρι 8. Αλλά πήρα και πολλά email από εκείνους που μας προειδοποιούν για τον κίνδυνο και λένε μα δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά. Στον, στο 118 αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίο δίπλωμα ευρυστεχνίας με τη δέουσα προστασία και αυτό δεν το κάνουμε τώρα. Άρα δηλαδή ε, θα πρέπει κανείς να βλέπει και τις δύο όψεις του νομίσματος και το δικό μας το καθήκον ως Κοινοβούλιο είναι να λάβουμε μια πολιτική απόφαση. Γι' αυτό λοιπόν εξακολουθώ να ισχυρίζουμε ότι αν το άρθρο θέλει πάση θυσία να ε, διαγράψει κάποια άρθρα, υπάρχουν στον κανονισμό κάποια άλλα, ε, διαγράψτε αυτά που δεν είναι σημαντικά. Αλλά όχι αυτά που είναι σημαντικά και το ξαναλέω λοιπόν το Κοινοβούλιο δεν επιτρέπεται να συμφωνήσει εδώ, γιατί αν το κάνει τότε θα παραβιάσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και αν το κάνει αυτό κάποιος άλλος θεσμός, αυτό είναι δική τους υπόθεση και δική τους ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν εμείς ε, να δεχόμεθα τις ευθύνες που μας μετακυλίουν άλλοι. Εμείς, ε, ε, η δουλειά μας είναι να εκπονούμε σωστό, δίκαιο και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εντάξει, θα τα ξανασκεφτούμε όλα αυτά, αλλά σας λέω για άλλη μια φορά με απόλυτη σαφήνεια. Εδώ δεν δόθηκε σήμερα το εναρκτήριο λάκτισμα για νέες διαπραγματεύσεις. Μα επουδενή. Μέχρι τώρα ισχύουν αυτά επί των οποίων έχουμε ε, διαπραγματευτεί και όλοι οι άλλοι που ε, λένε ότι πρέπει να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα τους λέω και εγώ ευχαριστώ πολύ, ε, συμφωνώ και επαυξάνω. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή, ε, ευχαριστούμε και όλους, ευχαριστούμε και τους ε, διερμηνείς γιατί ε, μας επέτρεψαν να ξεπεράσουμε κατά το χρόνο, κλείνει η συνεδρίαση. Έτσι κι αλλιώς το θέμα θα επανέλθει στην ημερήσια διάταξη και να σας επισημάνω ότι σήμερα το απόγευμα στις 3 η ώρα θα έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών για τρία μόνο λεπτά και μετά θα συνεχίσουμε με τις συνεδρίες και κλεισμένων των θυρών.